Πόσα μέλη είναι παρόντα άραγε. Λέω να αρχίσουμε αν, αν έχουν έρθει αρκετοί βουλευτές. Η κυρία Τούρινεν πάντως ήρθε. Λοιπόν, αν δεν απατώμε θα αρχίσουμε. Με το σημείο 17, πρώτη ανταλλαγή απόψεων, παρουσία εμπειροχνομόνων και εκπροσώπων ορισμένων εμπορικών εταίρων μας για την έκθεση της κυρίας Εμιλίας Τούρουνεν. Είναι έκθεση πρωτοβουλία για την πρόθεση τη πρόβαση των νέων στην αγορά εργασία, ενίσχυση του καθεστώτου τη άσκηση, τη πρακτική άσκηση και τη μαθητεία. Η κυρία εισηγήτρια παρακαλώ να έχει το λόγο για ολίγα λεπτά και μετά να αρχίσει η συζήτηση. Ύστερα δεν θα μιλήσουν και οι προσκεκλημένοι και προσκεκλημένες. Σας, ευχαριστώ. για τους νέους και τις ε, δυνατότητες που έχουν ε, οι νέοι ή μάλλον την έλλειψη των δυνατοτήτων που έχουν οι νέοι σε ό,τι αφορά την ε, κατάρτισή τους και την συμπερίληψή τους ή τον αποκλεισμό τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε το, την πρόκληση που υπάρχει πάνω από 5,5 εκατομμύρια νέων κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι. Υπάρχουν επίσης πολύ λίγες θέσεις μαθητευομένων. Τις οποίες, εντάξει, χρησιμοποιούμε. Ε, ουσιαστικά τους χρησιμοποιούμε ως ε, πάμφθινο εργατικό δυναμικό. Ξέρουμε ότι πάρα πολλοί νέοι φεύγουν από το εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς ουσιαστική κατάρτιση. Το θέμα είναι το γιατί. Γιατί οι νέοι αισθάνονται αποκλεισμένοι. Δεν είναι αρκετά ευέλικτοι. Άραγε. Αλλά ξέρουμε ότι το πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχει το ψυχολογικό πρόβλημα του αποκλεισμού και είναι λάθο τη Ευρωπαϊκή ένωση να δεχτεί κάτι τέτοιο. Επομένω, έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Για να την αντιμετωπίσουμε πρέπει να δράσουμε όμως. Πρέπει να αναλάβουμε τις πολιτικές μας ευθύνε. Και φυσικά και τα διάφορα κράτη πρέπει να αναλάβουν τις δικέ τους ευθύνε. Δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά. Θα ακούσουμε καλύτερα τους εμπειρογνώμονες που θα πούν καλύτερα που είναι πολύ ενδιαφέροντα άτομα από τα πανεπιστήμια, είναι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, είναι εκπρόσωποι των νέων, που μπορούν να μας εξηγήσουν πολύ καλύτερα την κατάσταση και το μέλλον για τους νέους. Πριν σας δώσω το λόγο, θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα Ερχόμαστε στο πρώτο τμήμα της ε, μήνυα ακρόασής μας, κατά τη διάρκεια του οποίου θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες. Κάνατε όλο αυτό το δρόμο να έρθετε εδώ πέρα και θα σας δώσω ακριβώς πέντε λεφτά γι' αυτό. Γιατί είμαστε με πολλούς προσκεκλημένους που θέλουν όλοι να λάβουν το λόγο. Κύριε Γιώργιο Μπρουνέλο, είσαστε στο τμήμα οικονομικών στην Πανεπιστήμιο της Παδούης. Για πέντε λεπτά θα σας δώσω το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω πολλά, αλλά λόγω της έλλειψης χρόνου θα πω λίγα. Λοιπόν, ποια είναι τα δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία στην αγορά εργασίας. Πρώτον, φεύγουν πολύ νωρίς από το σχολείο. Σε μερικές χώρες νέοι εργαζόμενοι παγιδεύονται σε προσωρινές εργασίες γιατί δεν έχουν επαρκή κατάρτιση. Βραχυπρόθεσμα σήμερα, μέσα στην κρίση, όποιος μπαίνει στην αγορά εργασίας μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ και μακροχρόνια προβλήματα χαμηλά εισοδήματα να υπάρξει ένα εφέ χαμένης γενιάς δηλαδή. Όπως έγινε στην Ιαπωνία τα τελευταία δέκα χρόνια και από το 90 ήδη γιατί η ανεργία αυξάνεται και είναι μακροχρόνια και η κρίση θα μειώσει ακόμα περαιτέρω τις θέσεις εργασίας. Δέστε τη Σουηδία, τη Φιλανδία και την Ιαπωνία πάλι. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να καταρτίζονται περισσότερο οι νέοι. Είναι εύκολο να το πούμε, δύσκολο να γίνει βέβαια. Αλλά οι οικονομολόγοι γνωρίζουν ότι είναι πολύ καλύτερο να δαπανηθούν χρήματα νωρίτερα στη ζωή για την κατάρτιση, ας πούμε, από την παιδική ηλικία ήδη, για την παιδεία. Γιατί αυτό αποδίδει στο μέλλον περισσότερο από άλλα άλλες μεθόδους. Και αν θέλουμε να έχουμε καλή μόρφωση πρέπει τα παιδιά να μένουν περισσότερο στο σχολείο. Άλλη πρόταση. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι αν αυξηθεί ο χρόνος της υποχρεωτικής παιδείας είναι καλύτερο το μέλλον των νέων. οι λιγότερο προνομιούχοι δεν θα μείνουν στο σχολείο παρά μόνο αν υποχρεωθούν βέβαια. Αυτό είναι σχέδιο δύσκολο να εφαρμοστεί, αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, επιδοτήσεις όπως στο ΙΤΑΒ. Οι επιδοτήσεις που δίνονται για την παιδεία σε παιδιά, σε νέους 16 ετών για να παραμείνουν στο σχολείο και έτσι να έχουν κάποια καλύτερα εισοδήματα. Αυτό φέρνει αποτελέσματα φαίνεται. Τώρα αν θέλουμε να παραμείνουν οι νέοι στα σχολεία περισσότερο πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό γίνεται ευκολότερα αν είναι πιο διαφοροποιημένο το σχολικό πρόγραμμα. Αν υπάρχει επαγγελματική κατάρτιση ας πούμε στο σχολείο. Αν το σχολικό σύστημα επιτρέπει τέτοια διαφοροποίηση είναι ευκολότερο τα παιδιά που θα ήθελαν να εγκαταλείψουν το σχολείο γιατί το βρίσκουν πολύ αφηρημένο να παραμείνουν. Τα πολύ αφηρημένα προγράμματα λοιπόν δεν ελκύουν τους νέους. Τώρα η πανεπιστημιακή μόρφωση. Ξέρουμε ότι σε περίπτωση κρίσης οι νέοι προσπαθούν να παραμείνουν στο πανεπιστήμιο γιατί ξέρουν ότι αν βγουν στην αγορά εργασίας θα έχουν πρόβλημα. Χαμηλά εισοδήματα, προσωρινή εργασία και θα ίσως να καταντήσουν χαμένη γενιά. Επομένω, Επομένως σε περιστάσεις κρίσης προτιμούν να παραμείνουν στο πανεπιστήμιο αλλά υπάρχουν έξοδα, έχουν κοστίζει η και μπορεί να φύγουν από το σχολείο και γι' αυτό. Θα ήταν εύκολο να σας πω εντάξει ας δαπανίσει περισσότερα η κυβέρνηση αλλά ξέρουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά, είναι άδεια τα ταμεία. Μειώνονται τα φορολογικά έσοδα, ζητούνται περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και εφόσον οι κυβερνήσεις κάνουν τέτοιες περικοπές πώς να ζητήσουμε περισσότερες δαπάνες. Το θέμα λοιπόν είναι Αφού στον ιδιωτικό τομέα πληρώνονται περισσότερο οι πιο καταρτισμένοι, θα μπορούσαν όσοι έχουν θέσεις που αμείβονται υψηλά να επιχορηγήσουν εκείνοι τους υπόμενους. Τέλος, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, η πολιτική για την παιδεία δείχνουν τα δεδομένα ότι δεν λειτουργεί για όσους τη χρειάζονται περισσότερο, για τους λιγότερο προνομιούχους. Χωρίς πολλές εξαιρέσεις μάλιστα. Υπάρχει ας πούμε το New Deal του ΙΤΑΒ για τους νέους. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, αλλά γενικότερα πρέπει η επαγγελματική κατάρτιση να συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό ή δίπλωμα και εδώ τελείωσα. Σας ευχαριστούμε για την αυτοπιταρχία που δείχνετε δίνω στον κύριο Τόμα Σβίκ από το Λουδοβίκιο Μαξιμίλιο Πανεπιστήμιο τη Μουνιχιλιάνιο. Πέντε λεπτά έχετε. Ε? Μαξιμιλιάνιο, ρε. Κύριος, θα μιλήσω για ένα διαφορετικό σύστημα το οποίο δεν αφορά τόσο τους νέους όπως έλεγε ο κύριος Μπρουνέλλο Ξέρουμε ότι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανεργία των νέων είναι μεγαλύτερη από τη η ανεργία των πιο ενήλικων, αλλά υπάρχουν πολλές ποικιλίε στην, ε, στον ποσοστό αυτό ανεργία σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δούμε τις πέντε χώρες που έχουν το υψηλότερο ρυθμό ανεργία σε ό,τι αφορά τους νέους, που είναι πολύ πιο υψηλό αυτός ο ρυθμός, Σουηδία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο και μια άλλη χώρα, οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από μια μικρότερη συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και αν τις συγκρίνουμε με άλλες χώρες που έχουν χαμηλή ανεργία όπως η Γερμανία, η Αυστρία, οι κάτω χώρες, η Σλοβενία κτλ. Οι χώρες αυτές έχουν υψηλότερο του μέσου όρου ε, ποσοστό μαθητείας και επαγγελματική κατάρτισης. Η μαθητεία οι μαθητεία λοιπόν, τα προγράμματα μαθητείας μπορούν να βοηθήσουν να μειωθεί η ανεργία των ε, νέων. Είναι το ερώτημα ή όχι. Εδώ τι μπορώ να πω. Μπορώ να πω ότι όταν εξετάσουμε την κατάσταση που επικρατεί στη Γερμανία, θα πρέπει να κάνουμε και κάποια σχόλια για τη στατιστική. Πρώτα απ' όλα. Στη Γερμανία πρέπει να πηγαίνει κανείς στο σχολείο μέχρι τα 18 και δεν μπορεί επομένως να πάρει επίδομα ανεργίας πριν από τα 18. Αν δούμε την ανεργία των νέων στη ηλικία των 22-23 χρονών ανεβαίνει εκθετικά η ενέργεια τους. Επιπλέον υπάρχουν πολλές επιλογές για να έχει κανείς ε, πλήρη σχολική <clears throat> απασχόληση. Υπάρχει το λεγόμενο σύστημα μετάβασης το οποίο κρατάει τους ανθρώπους μακριά από τις στατιστικές ανεργίες αλλά δεν τους δίνει κατά ένα εφαλτήριο σε ένα σύστημα μαθητείας το οποίο θα τους βοηθήσει να αποκομίσουν μετά κάποιες δεξιότητες στον χώρο εργασίας. Ούτε καν ένα ακαδημαϊκό δίπλωμα τους δίνει. Σε τέτοιους δύσκολους καιρούς το σύστημα μετάβασης διωγγώνεται και το βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι σαν ένα εναλλακτικό σύστημα, μένουν στο σχολείο παρά το γεγονό ότι δεν το θέλουν και φαίνεται ότι δεν είναι το πιο λογικό σύστημα λειτουργία. Απλώ κρατάει του νέου μακριά από την αγορά εργασία. Α πούμε ότι θέλουμε να δώσουμε τώρα επιδότηση στου εργοδότε για να έχουν περισσότερα προγράμματα μαθητεία. Αυτό φαίνεται να είναι δύσκολο να αυξήσουμε το ενδιαφέρον τους για τις μαθητείες. Γιατί το ποσοστό των, ε, της μαθητείας σε σχέση με τη συνολική εργατική δύναμη είναι σχετικά σταθερό. Αυξάνεται όταν είναι κρίση, μειώνεται όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αλλά το ποσοστό των ε, μαθητευομένων των τσιρακιών, όπως λέμε στη Γερμανία, είναι κάτι το οποίο είναι γενικά σταθερό και δεν αλλάζει τόσο εύκολα. Έχουμε διάφορα προγράμματα τα οποία έχουν σαν στόχο να παροτρύνουν τους εργοδότες να απασχολούν περισσότερο σε προγράμματα μαθητείας, αλλά δεν έχουν ευδοκιμήσει τόσο πολύ. αυτά τα προγράμματα. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί κανείς μόνο με επιδοτήσεις να παροτρύνει τις επιχειρήσεις να έχουν πιο πολλούς μαθητευόμενους. Εάν υπάρχει πραγματικά μια τέτοια ε, τάση, αυτό αφορά κυρίως τους ε, εργοδότες οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν μαθητευόμενους ως εναλλακτική και υπαλλακτική δύναμη για εκπαιδευμένους και μη εκπαιδευμένους εργαζομένους. Αλλά εδώ βλέπετε ότι η συνέπεια είναι ότι όταν τελειώσει η περίοδος μαθητείας δεν θα συνεχίσουν να εργάζονται οι μαθητευόμενοι και τελικά θα πάρουν μια εκπαίδευση χαμηλού επίπεδου, ιδίως στις χώρες αυτές όπου δεν υπάρχει διαδικασία πιστοποίησης ή σύστημα ελέγχου της ποιότητα των μαθητευομένων. Επομένως, ως εκ τούτου, μπορεί να είναι μαθητευόμενοι για 2-3 χρόνια, αλλά μετά θα μείνουν στον άσο, θα μείνουν εκτός αγοράς εργασίας, δεν θα έχουν ένα πιστοποιητικό υψηλής ποιότητας μαθητείας και τα άτομα αυτά θα έχουν ουσιαστικά πολλαπλές ουλές ως εργαζόμενοι και μέλη της αγοράς εργασίας. Δεν θα βρίσκουν εύκολα καλή δουλειά στο μέλλον. Και επομένω οι επιδοτήσεις αυτές δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι οι εργοδότες οι οποίοι προσλαμβάνουν άτομα που είναι σε μειονακτικές ομάδες πληθυσμού για να πάρουν ε, επιδοτήσεις δεν παίρνουν τον αντίστοιχο αριθμό μαθητιών οι εργοδότες εθίζονται στις επιδοτήσεις και γι' αυτό δεν παίρνουν πια μαθητευόμενους. Υπάρχει λοιπόν ένας πραγματικός κίνδυνος ότι ξεκινάει κανείς από τους μαθητευόμενους, μετά εθίζεται και τελικά κάνει μια συμβολή για τις ε, μαθητείες σε ένα περιορισμένο επίπεδο. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο αντιβαίνει στην ιδέα των επιδοτήσεων για τους εργοδότες οι οποίοι προσλαμβάνουν μαθητευόμενους. Και οδηγούμε έτσι ακόπως σε ορισμένες συστάσεις. Πιστεύω ότι τα μέτρα για την βελτίωση της ζήτηση στην αγορά εργασίας είναι και οι πιο αποτελεσματικές κινήσεις σε ό,τι αφορά και τους νέους. Δεν θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξω επιδοτήσει που είναι στοχευμένε σε μία ομάδα μονάχα, όπω είναι οι νέοι, τα άτομα που έχουν μειονεξία σε κάποιο επίπεδο. Αλλά όταν δημιουργεί κανεί μεγαλύτερη ζήτηση στον χώρο τη εργασία, εν γέννη και οι νέοι <clears throat> θα ευνοηθούν πέραν του μέσου όρου από όλου. Σα παρακαλώ να κλείσετε, λέει ο πρόεδρο. Η πρόεδρο, παρακαλώ να περατώσετε την παρέμβασή σα. Οι επιδοτήσεις λοιπόν θα πρέπει να έχουν σαν στόχο να μειώσουν και την ε, ανισότητα μεταξύ αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου και ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσει κανείς τα άτομα που έχουν ε, κάποια προβλήματα που είναι μειονεκτικά είναι με ειδικέ ενέργειες παροχή συμβουλών στα σχολεία πρωτού μπουν στην αγορά και όχι όταν μπουν στην αγορά εργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο τρίτο εμπειρογνώμων Κριστόφ μένγκ από το Ερευνητικό Κέντρο για την Εκπαίδευση και την Αγορά Εργασίας στο Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ. Πέντε λεπτά. Θα είμαι σύντομος. Και επί της ουσίας, όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές. Ε, ούτως ή άλλως με κάλυψαν σε κάποιο βαθμό. Δύο σημαντικά σχόλια έχω να κάνω. Καταρχάς, αυτούς που φεύγουν νωρίς το σχολείο και δεύτερον, αυτό που κατά την άποψή μου υπάρχει ένα πρόβλημα με την προσφορά ε, επαγγελματική κατάρτισης. Τι σημαίνει αυτό δεύτερο, ότι υπάρχει έτσι κάποιο πρόβλημα. Βλέπουμε ότι η μαθητεία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης είναι λιγότερες, λιγότερες δηλαδή θέσεις μαθητείας. Οι προηγούμενοι ομιλητέ είπαν ότι δεν είναι υπέρ των επιδοτήσεων. Οι περισσότερες, στις περισσότερες χώρες οι επαγγελματικές καταρτήσεις στην, στο χώρο εργασία, επιδοτούνται μέσω φόρων. Η άποψή μου είναι ότι οποιασδήποτε επιδοτήσεις δίνουμε σε επιχειρήσεις για τις μαθητείες θα πρέπει να τις αποσυνδέσουμε από το συγκυριακό οικονομικό κύκλο. Θα πρέπει να αυξήσουμε αντίθετα ε, στο, στις κακές ε, οικονομικές εποχές και στην, να τις μειώσουμε στις καλές, ούτως ώστε συνολικά να έχουμε κάποιες θέσεις μαθητείας. Αυτό ε, θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε ως σταθεροποιητή. Τη στιγμή που μπαίνουμε στην κρίση, δηλαδή, δεν είναι εκείνη η κατάλληλη στιγμή για τις επιδοτήσεις, για το αν θα αυξηθούν, ποιος θα τις πάρει κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας ήθικ των προτέρων που να λέει ότι όταν συμβεί αυτό, ας πούμε, στην οικονομία, την τάδε χρονική στιγμή, τότε αυξάνονται οι επιδοτήσεις, ας πούμε, για τη μαθητεία. Δεύτερον, η μείωση ε, των μαθητών που φεύγουν νωρίτερα από τα σχολεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μία από τις πρώτες προτεραιότητες στην ομιλία μου. Τα άτομα αυτά αποτελούν πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για τον εαυτό τους, γιατί δεν μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, αλλά έχουν πρόβλημα να ενταχθούν και στην κοινωνία. Και τελικά κοστίζουν λεφτά. Θα πρέπει να βρούμε μέτρα για να κρατήσουμε τα παιδιά στο σχολείο μέχρι να φτάσουν σε ένα επίπεδο εκπαιδευτικό που τους δίνει απαρκείς δεξιότητες και προσόντα για την αγορά εργασίας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι δύο μετρήσεις. Καταρχάς, ε, το σχολείο δεν θα πρέπει να είναι απλώς ένας τόπος που μαθαίνουν τα παιδιά. Είναι, μιλάμε για μια ομάδα μαθητών που έχουν πολλά και σύνθετα προβλήματα και το σχολείο πρέπει να βοηθήσει αυτά τα άτομα που φεύγουν όλοι από το σχολείο. Θα πρέπει να τα εντάξουμε στο σχολείο. Ε, και εκεί να μπουν οι κοινωνικοί λειτουργοί στο σχολείο για να βοηθήσουν τα παιδιά. Και όχι αργότερα. Δεύτερον, οι νέοι μας θα πρέπει να παίρνουν αποφάσεις σε νεαρή ηλικία. Πρέπει να πάρουν απόφαση τι είδους ε, μαθητεία, τι είδους σχολείο. Αλλά δεν είναι έτοιμοι ουσιαστικά να πάρουν τέτοιες αποφάσεις. Πολλά από τα άτομα που φεύγουν, φεύγουν από το σχολείο γιατί πήραν λάθος αποφάσεις. Νωρίς στη ζωή τους για το μέλλον τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, καθοδήγηση ε, ξανά και ξανά για τα παιδιά αυτά, ήδη από τα σχολεία, μέσω του σχολικού συστήματος. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι σε ποιο επίπεδο, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό χρειαζόμαστε κάποιες μετρήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποια είναι η κινητικότητα του, εργατικού συγγνώμη, δυναμικού και δεν ξέρουμε ποια είναι η κινητικότητα των νέων. Επομένως, χρειαζόμαστε τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπου τα σχολεία, οι επιχειρήσεις συνεργάζονται για να δώσουν την ε, επαγγελματική κατάρτιση και τα προσόντα που χρειάζονται τελικά οι επιχειρήσεις για να τους προσλάβουν. Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια με μετρήσει. και θα πρέπει με διάφορα μέτρα να προωθήσουμε ε, την κινητικότητα των νέων και να υποστηρίξουμε τα όσα γίνονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Τα μάλα, πρωτού στο επόμενο σημείο τη ημέρης τη διάταξη, να ακούσουμε αυτού οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο για να θέσουν ερωτήματα στου εμπειρογνώμονέ μα. Αυτό θα μα επιτρέψει να μην τα ανακατέψουμε όλα και να κάνουμε σούπα τα επιχειρήματα. Η κυρία θα ήθελε να μας εξηγήσει ίσως τι είναι αυτή η μάσκα που φορούσε, γιατί δεν είναι ακόμα προ... απόκριες, αλλά νομίζω ότι αφορά κάπως τους νέους οι οποίοι βρισκόνται σε επισφαλή θέση σχέση εργασίας. Η ιδέα είναι ότι όταν είναι κανείς νέος, μαθητευόμενος, τσιράκι, είναι ένα ανώνυμο ζώο, ένα άγνωστο ζώο, ένα ζώο που κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Επομένως, γι' αυτό το λόγο, αντί για σημαίες, αντί για μπαϊράκια, έχω αυτή τη μάσκα της αλληλεγγύης μαζί σας και επιτρέψτε μου να αφήσω αυτή τη μάσκα ενώπιον του μικροφόνου. Αν σας πειράζει θα τη βγάλω. Τη μάσκα δηλαδή. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν σε ερωτήσεις προς τους προσκεκλημένους μας. Καζά, Σταϊνμπρουκ, Μοράν, Ελμέρ και Σαρκά. Οι άλλοι συνάδελφοι θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την ε, θέση του στη συνέχεια τη συζήτηση. Θέλω να είμαι δυσάρεστη όπως πάντα και να σας δώσω το λόγο μόνο για δύο λεπτά στον καθένα. Γιατί έχουμε πολλούς προσκεκλημένους και προσκεκλημένες και πρέπει να κρατήσουμε το σωστό ρυθμό. Κύριε Κάζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να φύγω σύντομα γιατί στην Επιτροπή μου ψηφίζουν. Στην Οικονομική Επιτροπή και Οικονομική και Νομισματική. Και πρώτα και πάνω απ' όλα θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, την εισηγητή μάλλον, γιατί τη θαυμάσια εργασία της και την έκθεσή της που είναι ρεαλιστική. Ναι. Μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από αυτά τα οποία ελέγχθησαν από την εισηγήτρια, ο Σχιώδης και εγώ, εισηγητή. Κάποιε αλλαγέ όμω νομίζω θα ήταν χρήσιμε να τι υποδηλώσω. Είπε ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να αυξηθεί η χρηματοδότησή του. Αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ταμείο και με πιο αποδοτικό τρόπο. Γι' αυτό κατέθεσα και μία τροπολογία. Για αυτούς οι οποίοι φεύγουν πρόωρα από το σχολείο. Πιστεύω, μάλλον αυτοί που τελειώνουν το σχολείο ή φεύγουν από το σχολείο, θα πρέπει να έχουν επαγγελματική υποστήριξη και παροχή νουθεσιών για να μπορέσουν να βρουν δουλειά. Θα πρέπει να τους δώσουμε μια παροχή συμβουλών, ιδίω σε αυτού που φεύγουν πρόωρα από το σχολείο. Η παράγραφο αυτή που αναφέρεται στου πρόωρα αποχωρούντε από το σχολείο λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη στρατηγική του 2020 και όχι τη στρατηγική της Λισαβόνας. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αποδώσουμε μεγαλύτερη σημασία <clears throat> στη στρατηγική του 2020-2020 και όχι στη στρατηγική της Λισαβόνας που δεν επέτυχε τους επιδιωκόμενους στόχους. Περαιτέρω, θα πρέπει να αναφερθούμε και στην ανάγκη της οικονομικής ανεξαρτησίας για τους νέους ανθρώπους και να μην τους έχουμε εξαρτώμενους από κρατική αρρωγή και βοηθήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια σύνδεση όλων αυτών των ενεργειών με την διαβίου ε, εκπαίδευση και μαθητεία. Μια πολύ σημαντική ιδέα ήταν και η, εγγύηση, η ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους. Εγώ συμφωνώ με αυτή την πρωτοβουλία. Πιστεύω δε ότι μια ετήσια αξιολόγηση από την Κομισιόν ίσως είναι ιδιαίτερα επαχθής για την ίδια αυτή την Κομισιόν, αλλά κάθε δύο χρόνια θα είναι πολύ καλό να έχουμε μια αξιολόγηση από την πλευρά της Κομισιόν. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις που εγώ θέλω να κάνω. Τα κύρια θέματα που με ενδιαφέρουν. Η έκθεση είναι εξαιρετική. Δεν θέλω τώρα αυτή τη στιγμή να ζητήσω περαιτέρω αλλαγέ. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του εμπειρογνώμονε, των οποίων συμβολή ήταν αποφασιστική. θα τα ξαναπούμε πολλές φορές για την έκθεση του Βάνεν και τι τροπολογίε της, αλλά η επόμενη παρακαλώ να επικεντρώσει την προσοχή τους κυρίω σε ερωτήσεις προς του εμπειρογνώμονε, Η κυρία Σιλβάνα Ράπτη. Με συγχωρείτε κυρία Πρόεδρε που καθυστέρησα, αλλά είχα καλύψει και εγώ με τη μάσκα το μικρόφωνο και έπρεπε να το βγάλω. Ε, λοιπόν, ευχαριστώ την Έμιλη Τουρούνεν για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και νομίζω ότι πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι η σωστή εισηγήτρια για τη σωστή έκθεση. Γιατί θυμίζω ότι είναι το νεότερο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όχι μόνον αυτό προέρχεται από τη Δανία, μια χώρα που έχει καταφέρει να βελτιώσει πολύ τα πράγματα στην αγορά εργασίας για τους νέους. Άρα έχει να μας δώσει πολλά νέα στοιχεία, τα οποία βρίσκονται ήδη μέσα στην έκθεσή της. Για την έκθεση, όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στο χρονικό διάστημα που έρχεται μπροστά μας. Ε, την έκθεση θέλω να τη χαρακτηρίσω καταρχήν φιλόδοξη ελπιδοφόρα, με πολλές ευχές, αλλά από την άλλη πλευρά για να γίνουν αυτές οι ευχές πραγματικότητα νομίζω ότι θα πρέπει τις επόμενες εβδομάδες και μέχρι τις 31 Μαρτίου που έχουμε το όριο για τις τροπολογίες να μπορέσουμε να δώσουμε ε, πλαίσιο τέτοιο που να εφαρμοστούν κάποια πράγματα. Παράδειγμα, το σημείο 18 και το θέμα της εγγύησης. Θα πρέπει να το διατυπώσουμε με ένα τέτοιο τρόπο και νομίζω ότι μπορούμε όλοι μαζί να σκεφτούμε και να βοηθήσουμε, ώστε πραγματικά να βοηθήσουμε τους νέους. Δεν θα ασχοληθώ άλλο με το περιεχόμενο της έκθεσης, αλλά ακούγοντας με πολύ προσοχή τους τρεις εμπειρογνώμονες, σχημάτισα την εντύπωση ότι όλα τα πράγματα είναι η παιδεία όλα τα πράγματα, όλη η βάση βρίσκεται στην εκπαίδευση. Είναι λιγάκι σαν την υγεία. Είναι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε. Είναι καλύτερα να δίνουμε χρήματα και α, μέρημνα στην αρχή του σχολικού βίου, στην αρχή της σχολικής ζωής, ώστε να μπορούμε μετά πραγματικά να μην έχουμε προβλήματα ή να έχουμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Όσον αφορά την κατάρτιση, θα ήθελα να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες και περιμένω έτσι με πολύ ανυπομονησία τη γνώμη τους. Η κατάρτιση δεν θα πρέπει να είναι στοχευμένη σε τομείς που πραγματικά χρειάζεται η κοινωνία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι τα στάζ και η μαθητεία. Ε, μιλήσατε για επιδότηση. Έχω την αίσθηση... Ah, ε, Έχω την αίσθηση ότι τα στάζ είναι μια ασπιρίνη για την ανεργία. Οι ασπιρίνες είναι καλές για λίγο, δεν μπορούν όμως να διαρκούν πολύ. Και κλείνοντας, νομίζω ότι η μαθητεία θα πρέπει πάντοτε να είναι αμοιβόμενη, έστω και συμβολικά. Μέχρι Madame ε, Κυρία Στάινμπρουκ και μετά η κυρία Μορέν. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Ράπτη, δηλαδή το θέμα της μαθητείας και θα ήθελα να έχω την άποψη των ε, εμπειρογνωμόνων για αυτό το θέμα, αλλά προηγουμένως δεν θα ήθελα να παραλείψω να αναφέρω τα προβλήματα των μαθητευομένων στην Ευρώπη εν γέννη. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει όλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άμα δω την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξέρω ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός μάθητευομένων οι οποίοι μένουν εδώ για λίγους μήνες μονάχα. Είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερα τους νέους αυτούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, εκεί πρέπει να έχουμε κι εμείς βέλτιστες πρακτικές ως βουλευτές, να δίνουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες μαθητείας σε αυτούς, ώστε τα άτομα αυτά να βοηθηθούν για τη συνέχιση της ε, καριέρας τους, να βρουν θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν κάποια αξιοπρέπεια και όχι να τους βάζουμε σε μειονεκτική θέση. Είναι χρήσιμο λοιπόν να υπάρχει το σωστό πλαίσιο μαθητείας, γι' αυτό κάνω και αυτή την έκκληση και προς τη δείξη του Κοινοβουλίου να υπάρχει η απαραίτητη ε, παροχή υπηρεσιών προς τους μαθητευόμενους, ιδίως όταν αυτή είναι άμυστη. Ο κύριος Έλμερ, Μωρέν. Μωγά. Κυρία Μωγά, άκουσα τους τρεις εμπειρογνώμονες και νομίζω ότι το πρώτο θέμα που πρέπει να θέσουμε όλοι μαζί είναι τι νόημα θέλουμε να δώσουμε στο σχολείο. Το σχολείο δημιουργείται για να συγκρατήσει τους νέους ε, στο σχολείο, να τους κρατήσει εκεί ε, παρά τη θέλησή τους, να τους δώσει κάποια εφόδια ε, μέχρι να βγουν στην αγορά εργασίας ή για να τους διαμορφώσει, να τους δώσει ένα επίπεδο διπλώματος που θα τους ανοίξει συνεχεία τις πόρτες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό χώρο ζωής και εργασίας χωρίς το σχολείο να παίξει αυτόν τον πρώτο ρόλο, αυτόν τον πρωταρχικό ρόλο. Να έρθουμε λοιπόν στην ουσία του σχολείου. Το σχολείο δεν είναι εκεί για να φυλακίσει τους νέους, αλλά για να τους διαμορφώσει μέχρι το πτυχίο τους. Δεύτερον, ε, αυτοί που φεύγουν το σχολείο χωρίς προσόντα. Είναι ένα πρόβλημα τεράστιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο το να έχουμε μια τέτοια μάζα νέων που βγαίνουν από το σχολείο και δεν έχουν τίποτα στα χέρια τους, χωρίς προσόντα. Ακούσαμε τους εμπειρογνώμονες να μας λένε ότι θα πρέπει η κοινωνική λειτουργία να πάνε ήδη στο σχολείο για να βοηθήσουν τα παιδιά, ε, ούτως ώστε να μειωθούν ε, αυτοί που φεύγουν νωρίς από το σχολείο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά τους εξατομικευμένα και θα πρέπει τους ανθρώπους αυτούς που ασχολούνται με την επαγγελματική κατάσταση στο σχολείο, να τους συνδέσουμε με διάφορα δίκτυα στο εξωτερικό για να ενημερώσουν πραγματικά και να πλαισιώσουν τους νέου ε, και να τους κατευθύνουν και προ τη μαθητή αν χρειάζεται. Επομένω, υπάρχει ένα, υπάρχει ένα θέμα το πρόωρα αποχωρούνται από το σχολείο, θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ ε, σοβαρά. Τρίτο σημείο είναι η μαθητεία, το στάζ. Έπειτα, διαφορετικά μέτρα για να περάσουμε από το χώρο της κατάρτισης στο χώρο της εργασίας. Δηλαδή η εναλλαγή από το χώρο της κατάρτισης στο χώρο της εργασίας. Προσοχή για όλους. Οι νέοι έχουν δυσκολίες να βρουν καταρχάς ανθρώπους που θα τους δώσουν μαθητείες, να, να βρουν στάζ. Είναι τεράστια αυτή η δυσκολία που έχουν. Ε, το ξέρουμε και εμεί οι ίδιοι, γιατί κάποια στιγμή χρειάστηκε να σπρώξουμε για να πάρει κάποιο νέο ε, μια θέση μαθητεία. Αυτή η δυσκολία προέρχεται από το γεγονό ότι για να είναι αποτελεσματικό το στάζ και η μαθητεία θα πρέπει να υπάρχει ένα υπεύθυνο. Θα πρέπει να υπάρχει στην ε, επιχείρηση, στο χώρο που υποδέχεται του νέου, σε ένα ας πούμε βοηθό, ε, ένα άνθρωπο ο οποίο πλαισιώνει τον νέο, που τον βοηθάει, ένα διδάσκαλο αν θέλετε. Τώρα ο κύριος Έλμερ και μετά ο κύριος Θωμάς Μαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από όλα όσα ακούσαμε μέχρι τώρα, τονίστηκε η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Φυσικά είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Αλλά οι λύσεις που προτείνονται ήταν όλες υποχρεωτικές ας πούμε την ηλικία κατά την οποία έχει κανείς το δικαίωμα να φύγει από το σχολείο και τέτοια και όλο και περισσότερο και περισσότερες κυβερνητικές δαπάνες. Από κοινική απόψεως θα έλεγε κανείς ότι απλώς προσπαθούν να κρατήσουν τους νέους έξω από τους καταλόγους των ανέργων για να τους κρατήσουν στο σχολείο μόνο και μόνο γι' αυτό. Αλλά δεν σκεφτήκαμε καθόλου ποια είναι η ζήτηση που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Δεν είναι βέβαιο ότι αν έχουν κατάλληλη κατάρτιση οι νέοι θα έχουν και δουλειές, Άμα δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, όσοι κατάρτιση και να έχουν όσοι βγαίνουν από το σχολείο νωρί ή αργά, θα καταλήξουν άνεργοι και άνεργες. Άρα πρέπει να δούμε και την πλευρά της ζήτησης, διότι οι επιχειρήσεις επενδύουν είτε σε υλικά είτε σε εργαζόμενους, μόνο εάν έχουν την προοπτική ανάπτυξης και κερδών. Και γι' αυτό το να σκεφτόμαστε όλο υποχρεωτικά μέτρα, περισσότερες δαπάνες, δεν είναι σίγουρο ότι είναι αυτό που πρέπει να τονίσουμε. Καλύτερο θα ήταν να τονώσουμε την οικονομία. Γιατί έτσι θα αυξηθεί από μόνο του το επίπεδο της απασχόλησης. Λυπούμε αν σας ε, αν καθίσταμε βαρετός γιατί αυτά τα έχω πει πολλές φορές αν υπήρχαν λιγότεροι φόροι και λιγότερη νομοθεσία θα υπήρχε μεγαλύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη απασχόληση καθώς και λιγότεροι άνεργοι και άνεργες. Ευχαριστούμε κύριε Έλμερ. Δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να συμφωνήσει μαζί σας αλλά η επικοινωνία είναι πολλές φορές η τέχνη της επανάληψης. Είναι αναγκαίο να περνάει κανείς τις ιδέες. Τόμας Μαν και μετά Φέρκας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα θέμα το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό που είναι αυτοί οι οποίοι φεύγουν πρόωρα από το σχολείο. Πάρα πολλά άτομα βαριούνται στο σχολείο γιατί δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα με την παιδεία την οποία παίρνουν στο σχολείο. Πολλοί δεν έχουν και πρακτικές δεν έχουν πρακτικά ταλέντα τα οποία μπορούν να αποκομίσουν από όλα αυτά και αυτά τα άτομα επομένω δεν προχωρούν με τη σχολική εκπαίδευση. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχουμε ένα καλό παράδειγμα για το πώ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να βοηθήσει αυτά τα άτομα, να δώσει τα άτομα αυτά <clears throat> σε αυτού που στη Γερμανία παραγωγικά δεν παίρνουν κανένα απολυτήριο γυμνασίου ή αντίστοιχου σχολείου. Να έχουν τη δυνατότητα σε μικρέ ομάδε να μάθουν μια τέχνη. Να έχουμε λοιπόν ένα μικρό αριθμό ε, μαθητών που θα μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο. Πολλές φορές αυτοί οι οποίοι είναι οι νέοι που είναι οι μόνοι οι οποίοι σηκώνται το πρωί και έχουν κάτι να κάνουν γιατί η υπόλοιπη οικογένεια είναι άνεργη, πηγαίνουν σε μια επιχείρηση, έχουν μια εμπειρία η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη για αυτούς γιατί καταλαβαίνουν ότι κάποιο τους χρειάζεται, έχουν κάποια προσόντα τα οποία τα εκτιμά η αγορά και θεωρούν για πρώτη φορά στη ζωή τους ότι μπορούν να κάνουν κάποια πρόοδο. Αυτό τους δίνει αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περαιτέρω καριέρα τους. Για αυτά τα άτομα λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε, να κάνουμε με τον τρόπο αυτό εξοικονόμηση από όλες τις άλλες διορθωτικές επενδύσεις οι οποίες δεν λύνουν το πρόβλημα. Θα πρέπει εκεί ακριβώς να δώσουμε την έμφαση, να βοηθήσουμε αυτά τα συγκεκριμένα άτομα και κάνουμε μεγάλες προσπάθειες να έχουμε κατάρτιση σε εθνικό επίπεδο, γιατί εκεί θα πρέπει να δοθεί η έμφαση, εκεί πέρα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα, να τα κινητοποιήσουμε, να του δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τι ευκαιρίε. Έτσι η Ευρώπη θα μπορούσε να δώσει πολύ καλά παραδείγματα για όλου. Δυστυχώ πρέπει να πάω τώρα σε μια άλλη επιτροπή, γιατί ψηφίζουν εκεί. Αλλά δύο από του συνεργάτε μου είναι εδώ και θα καταγράψουν όλα αυτά τα οποία θα πείτε ω εμπειρογνώμονε και ω συνάδελφοι και σα ευχαριστώ εξ αρχή. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Θέρκας και μετά στην κυρία Τουρούνεν για να τεθούν και ερωτήματα από όλους σας τους ε, εμπειρογνώμους. Κύριος Θέρκας. Πρόεδρε, είναι προφανές ότι το θέμα της κατάρτισης, ο τομέας κατάρτισης είναι ο πλέον βασικός για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των, της ανεργίας των νέων. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου έχουμε τρομερά νούμερα ανεργίας ε, και παρόλα αυτά ε, οι νέοι λαμβάνουν ε, εκπαίδευση. αλλά δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες αγοράς εργασίας. Έχουμε τρομερά, τρομές αποτυχίες στο σχολείο και παρόλα αυτά βέβαια έχουμε και πολύ, πάρα πολλούς φοιτητέ, περισσότερους από όσους χρειαζόμαστε. Και τελικά έχουμε πάρα πολλές τρύπες στην αγορά εργασίας που καλύπτονται από μετανάστες. Υπάρχει κατάρτιση, υπάρχει εκπαίδευση, αλλά γίνεται με διαφορετικό τρόπο σε άλλο χώρο, σε άλλους τομείς από αυτό που ζητάει η αγορά εργασίας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ε, να αναλύσουμε τις πληροφορίες. Γιατί οι πληροφορίες αυτές ε, μας εξηγούν ε, τις αποτυχίες ε, των νέων στο εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μου. Ε, οι εμπειρογνώμονες μίλησαν για αυτό το ευαίσθητο τμήμα του πληθυσμού. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι όταν επιδεινώνονται οι βιομηχανικές σχέσεις, όταν υπάρχει πρόβλημα με, την, με τις θέσεις εργασίας, την πληρώνουν πρώτα οι πιο ευαίσθητοι νέοι. Πάντα είναι, οι νέοι είναι τα θύματα. Πώς μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να βρούμε τρόπους ε, και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκεί όπου γεννάται, δηλαδή εκεί που στο επίπεδο όπου δημιουργούνται προβλήματα για τους νέους. Γιατί είναι τόσο ευαίσθητοι, γιατί είναι τόσο εκτεθειμένοι. Η παράγραφος F λέει ότι στη Δανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, η, η, πέτη για τα προβλήματα των ε, νέων είναι η, τα ελάχιστα εισοδήματα. Είναι λάθος αυτό. Είναι σωστό. Ε, το να εγγυόμαστε τα, τα ελάχιστα εισοδήματα είναι κακό δηλαδή και δημιουργεί προβλήματα. Ε, Σας ευχαριστούμε. Κυρία Τουρούνεν έχει το λόγο. Φοβάμαι ότι δεν είναι σφάλμα μετάφρασης. Μα θα έχετε, μπορείτε να συγκεντρωθείτε λιγάκι στα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να θέσετε. Θα ξαναγυρίσω με τον κύριο Σέρκας στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ εμπειρογνώμονες που ήρθατε εδώ και δώσατε αυτές τις τόσο σαφείς και συγκεκριμένες παρουσιάσεις. Ένα, ένα ερώτημα. Ένα ή περισσότερα, περισσότερα μάλλον. Το πρώτο από τα περισσότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ μαθητείας και Τη της του ασκουμένου με την κατάσταση του μαθητευόμενου. Υπάρχει έλλειψη μαθητιών, αλλά υπάρχουν πολλές θέσεις ασκουμένων που αντικαθιστούν τις πραγματικές θέσεις εργασίας. Ίσως θέλετε να σχολιάσετε αυτό το γεγονός. Δεύτερον, είπατε ότι η παιδεία είναι το πραγματικό εφαλτήριο για την αγορά εργασίας. Συμφωνώ. Αλλά τι άλλο μπορείτε να δείτε για τη δεύτερη φάση όταν έχει κανείς πολύ καλή παιδεία, μεν, και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Χέλμερ, βλέπετε όλα αυτά τα άτομα τα οποία είναι υψηλοπροσοντούχα να πουλάνε, να φτιάχνουν χάμπουργκες στο McDonald's. Λέτε επίσης ότι θα πρέπει να επιδοτούμε τους εργοδότες ή πρέπει να τους υποχρεώνουμε να παίρνουν μαθητευόμενους. Ποια είναι η πρότασή σας. Τέλος είπατε ότι στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο μπορούμε πράγματι να εξασφαλίσουμε την απασχόληση και λέτε ότι θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υποστηρίξουμε τι τοπικέ και περιφερειακέ πρωτοβουλίε. Τι είδου πρωτοβουλίε είναι αυτέ όμω που θέλετε να υποστηρίξετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάλι θα δώσω το λόγο σε καθένα από του εμπειρογνώμονε για δύο λεπτά και ξεκινώ από τον καθηγητή Γιώργιο Μπουνέλο. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει. Φυσικά δεν μπορώ να απαντήσω σε όλε τι ερωτήσει. Ένα σχόλιο για την εκπαίδευση. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι κατά μέσο όρο, όσο περισσότερο εκπαιδευμένος είναι κανεί τόσο περισσότερο πιθανό είναι να βρει μια δουλειά. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι η πιθανότητα ανεργία είναι μηδενική. Αλλά αν είσαι καλύτερα εκπαιδευμένο, θα πάρεις, ακόμη και αν είσαι είτε νέος είτε ενήλικας, ε, είναι πιο πιθανό να περάσεις στο επόμενο στάδιο. Δεν λέω ότι η υπερβολική εκπαίδευση δεν είναι και αυτή πρόβλημα. Τώρα, για την προσφορά. Από τα στοιχεία που έχουμε, φαίνεται ότι αν η Ευρώπη ανοίξει περισσότερο την αγορά στον ανταγωνισμό, αυτό θα μειώσει την απασχόληση και την κατάρτιση. Ε, επίσης είμαι σκεπτικιστής για τις επιδοτήσεις για τη μαθητεία, γιατί από τα στοιχεία που έχουμε δεν δείχνουν, δεν φαίνεται ότι λειτουργούν. Ίσως λοιπόν ε, οι μακροοικονομικές πολιτικές θα ήταν μια καλή εναλλακτική λύση. Ε, Ευχαριστώ. Ο καθηγητής Τόμας Σφίγγ. Υπήρχε μια, μια ερώτηση για τα θέματα της ε, επιδότησης. Προφανώς, αν υποχρεώσουμε τους εργοδότες να παίρνουν τσιράκι, αυτό δεν θα είναι θετικό. Καλύτερο θα είναι να πείσουμε τους νέους να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση πρώτα και μετά θα έχουν καλύτερη ευκαιρία να βρουν μια κατάλληλη θέση μαθητείας. Γιατί δεν πάει κανείς μακριά με το να υποχρεώνει με το ζόρι τους εργοδότες να παίρνουν μαθητε, μαθητευόμενους. Και βλέπετε ότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης. Τα γοριά γίνονται μηχανικοί αυτοκινήτων, τα κορίτσια γίνονται κομμότριες, γιατί αυτό νομίζουν ότι είναι η μόνη μορφή μαθητείας η οποία είναι χρήσιμη για αυτούς. Χρειάζεται λοιπόν παροχή συμβουλών και πληροφόρηση να ξέρουν ποιε είναι όλες οι δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους και να έρθουν πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες. Υπάρχουν σχολεία τα οποία έχουν μια πραγματικά θετική και ενεργητική προσέγγιση στους τοπικούς εργοδότες για να εξηγήσουν σε τι μπορούν να βοηθήσουν οι μαθητευόμενοι και αυτό είναι πιο αποτελεσματικό από το να έχουμε επιδοτήσει να υποχρεώνουμε με το στανιό του εργοδότε να προσλαμβάνουν μαθητευόμενοι. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρο. Κύριο ναι. Μέγγε. Το πρώτο ερώτημα το οποίο απευθύνθηκε σε μένα νομίζω ότι προέρχεται από το γεγονό ότι εγώ μίλησα για τοπικέ και περιφερειακέ πρωτοβουλίε και το ερώτημα τι μπορεί να γίνει αυτό από τα κράτη-μέλη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μα είναι ότι παρά το γεγονό ότι πρέπει να ξεκινήσουμε στο τοπικό περιφερειακό επίπεδο, γιατί εκεί είναι που οι εταιρείε και τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα. Πέραν αυτού βέβαια πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε οικονομικού τομεί οι οποίοι λειτουργούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Βέβαια, η οικονομική κρίση χτυπάει τα περιφερειακά επίπεδα διαφορετικά, γιατί επηρεάζει διαφορετικά τους οικονομικούς τομείς. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο είναι η υποστήριξη, η οποία θα υποστηρίξει τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε οικονομική κάμψη, γιατί θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι παρόλα αυτά θα εξακολουθούν να υπάρχουν διαδικασίες μαθητείας ακόμα και σε περιοχές στην Κάμψη. Κάτι άλλο που θέλω να πω σε σχέση με τις αντικυκλικού χαρακτήρα επιδοτήσεις για μαθητεία. Θα πρέπει να είμαστε σαφέστατοι στο να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ αυτών που πρέπει να επιδοτήσουμε και αυτές που, αυτών που δεν πρέπει να παίρνουν επιδοτήσεις. Κατά τη δική μου άποψη, σε καιρό ύφεση, οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να πάρουν επιδοτήσεις είναι αυτές σε οικονομικούς τομείς που έχουν καλές μελλοντικέ προοπτικές. Αλλιώς ο κίνδυνο είναι ότι επιδοτούμε μαθητές σε οικονομικούς τομείς οι οποίοι δεν έχουν μέλλον, δεν έχουν οικονομικές προοπτικές και εκπαιδεύουμε άτομα για θέσει εργασίας οι οποίες θα εξαφανιστούν έτσι κι αλλιώς μέσα στην επόμενη δεκαετία. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να κάνουμε τη διαφοροποίηση μεταξύ ασκουμένων και μαθητευομένων. Οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να κάνουν μακροχρόνιες διαδικασίες μαθητείας με κατάρτιση παράλληλη, με σαφή διπλώματα στο τέλος που βοηθούν τους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας. Οι θέσεις ασκουμένων είναι για αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν κάνει μια εκπαιδευτική πορεία η οποία τους έφερε σε ένα καλό επίπεδο αλλά στη συνέχεια θέλουν να αποκομίσουν εμπειρία σε επίπεδο εργασίας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει ποτέ τις μαθητείες. Δεύτερο τμήμα. Πάμε στο δεύτερο τμήμα αυτής ακρόασης και από τους κοινωνικούς εταίρους θα δώσω το λόγο αλφαβητικά στη Julian Beer από το ETUC. Πέντε λεφτά. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Πριν ε, σας δώσω την άποψη της ETUC, θέλω να χαιρετήσω την πρωτοβουλία αυτής της έκθεσης που θέτει ένα ουσιαστικό θέμα για τους νέους Ευρωπαίους και μια ουσιαστική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ερώτηση αυτή είναι το πρώτο μέλημα των νέων της Ευρώπης και δεν είναι καινούριο. Ας ε, θυμηθούμε το, τη σφιγμομέτρηση του Ευρωβαρόμετρου του 2002, εγώ συμμετείχα σε αυτή. Ε, η σφιγμομέτρηση αυτή έλεγε ότι η απασχόληση και η καταπολέμηση της ανεργίας είναι η πρώτη ε, ανησυχία των νέων πριν από τη δημοκρατία και όλα τα υπόλοιπα. Ποια είναι η προσέγγιση των νέων σήμερα. Θέλουν να ζήσουν ε, τη ζωή τους, να έχουν μια ποιοτική δουλειά, θέλουν να έχουν μια τα είπαμε το κεφάλι τους. Οι νέοι είναι ιδιαίτερα ευπαθείς, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε αυτή την περίοδο όπου η απασχόληση είναι ασταθής. Γνωρίζουμε το πλαίσιο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ε, τα ποσοστά ανεργίας το δείχνουν ε, και η έκθεση το δείχνει ανάκληφα. Για τους νέους Ευρωπαίους που έχουν την ευκαιρία εντό αγωγικών να έχουν μια θέση απασχόλησης, αυτή η απασχόληση δεν είναι παρόλα αυτά Για τα δύο τρίτα των νέων της Ευρώπης σήμερα ε, ε, η δουλειά σημαίνει ε, μερική απασχόληση, εποχιακή απασχόληση, έκτακτη απασχόληση ή αδήλωτη απασχόληση. Αυτές οι θέσεις ε, συνοδεύονται με χαμηλούς μισθούς, δύσκολες, συνθήκε, συνθήκες, έλλειψη κατάρτισης, προβλήματα στην κοινωνική προστασία και στην προοπτική για την καριέρα. Δεν είναι εύκολο λοιπόν μέσα σαν να θυμηθούμε ότι το δικαίωμα για σύμβαση αορίστου χρόνου θα πρέπει να είναι ο κανόνας, ενώ θεωρείται τελικά προνόμιο. Αυτή η κατάσταση φυσικά έχει συνέπειε στην καθημερινότητα των νέων, το είπαν κάποιοι, ε, εξάρτηση από το κράτο, αλλά και από του γονεί. Και από του παππούδε ακόμα. Ε, συχνά ε, ζουν μέχρι πολύ μεγάλη, μέχρι προχωρημένη ηλικία με τους γονεί και τους παππούδες, γιατί δεν έχουν ε, τη δυνατότητα να πληρώσουν τη δική του στέγη. Ε, τελικά, ποιο είναι το μήνυμα το συνεταιριστικό τη ETUC. Όταν μιλάμε για την απασχόληση των νέων, το, το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ποιότητα της ε, θέσης απασχόλησης των νέων. Οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας θα πρέπει να συνοδευτούν από τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων. Θα πρέπει να προλάβουν οποιοδήποτε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων αντίον των νέων. Ε, σε αυτό το πλαίσιο εμείς η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θεωρούμε ότι η ασφάλεια είναι ένας δρόμος ε, που πρέπει να διερευνήσουμε, ε, αλλά είναι επικίνδυνος και δεν είναι προσαρμοσμένος ε, στα δεδομένα. όλα σας είπα, όλα σας είπα δείχνουν, απαριθμούν μάλλον τις δυσκολίες που έχουν οι νέοι. Νομίζω ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια πάνω απ' όλα για να εξισορροπήσουμε την δουλειά με τον τρόπο ζωής. Επίσης, ε, τα μέτρα και οι πολιτικές θα πρέπει να συνοδεύουν η μία, τα μεν δε και παράλληλα να υπάρχει μόνιμος διάλογος με τα συνδικάτα και τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων. Η έκθεση λέει ότι η πρωτοβουλία ε, Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Νεότητα δεν θα πρέπει να μείνουν και γράμματα καινού περιεχομένου. Ε, τι γίνεται το, με την εφαρμογή του. Θα πρέπει να ρωτήσουμε και τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να αποφύγουμε την ανεργία ε, μακράς διάρκειας μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Επίσης, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα ε, σε όλες τις κυβερνήσεις για να υπάρχει ε, εκπαίδευση ποιότητας, ανοιχτή σε όλους τους ε, πολίτες, ανεξάρτητα από την θρησκεία τους, την προέλευσή τους, την κοινωνική και την φυλή τους. Θα πρέπει λοιπόν η κατάρτιση και εκπαίδευση να είναι προσαρμοσμένη και το δίπλωμα είναι το καλύτερο εχέγγυο απέναντι στην ανεργία. Οι νέοι πριν επιλέξουν οποιαδήποτε καριέρα θα πρέπει να γνωρίζουν τι προοπτικές υπάρχουν, αν θα έχουν δουλειά ή όχι και ποια είναι τα ποσοστά, να, τι δυνατότητες έχουν να βρουν δουλειά. Και βεβαίως, επειδή μιλήσατε για το θέμα της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου, δεν θα πω άλλα πράγματα, είναι πολύ σημαντικό όμως. Δύο τελευταία σημεία. Να σας ενημερώσω στα πλαίσια της ε, εκστρατείας του 2010 για ένα New Deal για τα κοινωνικά θέματα, θέλουμε να υπάρχει και μια εγγύηση για τους νέους, ε, εκπαίδευση, κατάρτιση, ποιοτική θέση απασχόλησης, ε, μαζί με μέτρα για την ε, προσληψιμότητα των νέων. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε στην διάσκεψη στη Μαδρίτη τέλος Απριλίου, που το θέμα της είναι νέοι και απασχόληση. Επίσης, το να στοιχηματίσουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Νεολαία δεν πρέπει να είναι κίνδυνο, αλλά εγγύηση για την Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Εξ ονόματο του Business Europe, ο κύριος Μάθιου Φίγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ, να σας συγχαρώ για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Είναι, όπως είπαν και άλλοι, ένα μακροχρόνιο δομικό πρόβλημα η ανεργία των νέων που έχει χειροτερέψει πολύ από την κρίση. Και οι Ευρωπαίοι εργοδότες θεωρούν ότι χρειάζεται μεγάλη ανάλυση και σκέψη για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να μην χαθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα αλλά και να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου όλες οι δεξιότητες των νέων δεν χρησιμοποιούνται. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο θα τονίσω ιδιαίτερα δύο θέματα και θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω μερικά πράγματα που είπαν άλλοι. Ο εξυγχρονισμός των συστημάτων της παιδείας και η διοργάνωση της αγοράς εργασίας. Πριν πισέλθω σε αυτά, μερικές παρατηρήσεις για τη στρατηγική του 2020 και μετά. Εμείς ε, δεχόμαστε τις προτεραιότητες και τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη εκφραστεί εδώ, δεν είναι βέβαια καινούργιε, αλλά χρειάζεται κάποια νέα ορμή, κάποια καινοτομία στην κατάρτιση των νέων, ιδιαίτερα εκείνων που μετακινούνται πολύ, που αρχίζουν την επαγγελματική του καριέρα. Η στρατηγική αυτή για την Ευρώπη το 2020 και μετά είναι κάτι που πρέπει επιγόντως να λυθεί ιδιαίτερα ως προς τα θέματα της αγοράς εργασίας και της κατάρτισης. Ε, εμείς στο Business Europe έχουμε τελευταία κάνει ένα δημοσίευμα Growth for Growth όπου δηλώνουμε ρητά ότι οι ποιες είναι οι προτεραιότητες μας για την ανάπτυξη και θεωρούμε ότι αν από το 1 αυξηθεί στο 2% η δυνατότητά μας ανάπτυξης, αυτό από μόνο του θα αυξήσει κατά 6,5% τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Και εφόσον διορθωθεί η κατάσταση της ανεργίας, τότε το 2020 θα μπορούσαμε να τονίσουμε και το θέμα των ολοκληρωμένη της ολοκληρωμένης αγοράς εργασίας με τις συμφωνίες πλαίσια που θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα. Αυτό δείχνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να βρουν εξισορροπημένες λύσεις για να μην ε, μειωθεί η ανάπτυξη. Επίσης, αν λάβουμε υπόψη μας και τα δημογραφικά, δηλαδή τη γύρανση του πληθυσμού, πρέπει η αγορά εργασίας να αναπτυχθεί γιατί δεν μπορούμε πια να δεχτούμε ότι οι ίδιες ομάδες εργαζομένων θα παραμένουν αιωνίως στην αγορά εργασίας. Για να μην επαναλάβω αυτά που είπαν προηγούμενοι για την κατάρτιση, θα έλεγα ότι το θέμα αυτό αφορά το κατά πόσον συνδυάζονται οι καταρτήσεις με την προσφορά στην αγορά εργασίας ή τη ζήτηση. Ο εξυγχρονισμός των εκπαιδευτικών συστημάτων για την προετοιμασία των νέων για την πρώτη τους δουλειά σημαίνει ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο μέσα στην παιδεία. Η επιχείρηση είναι ο καλύτερος τόπος μετάδοσης των πληροφοριών για τις ανάγκες που πραγματικά υπάρχουν και έτσι την προετοιμασία των προτιμήσεων των νέων για κατάρτιση, για να ανταποκρίνονται οι καταρτήσεις στις αλλαγές της αγοράς εργασίας. Στο έχει γίνει μια πρόβλεψη ότι μεταξύ των 80 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας που θα υπάρξουν μέχρι το 2020 οι περισσότερες θα απαιτούν υψηλή κατάρτιση και δεξιότητες. Γιατί οι κενές θέσεις που υπάρχουν σε πολλές χώρες μέλη όπου σημειώνεται και ανεργία παράλληλα 800.000 ας πούμε τέτοιες κενές θέσεις στη Γερμανία σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Και αυτό πρέπει να διορθωθεί από το εκπαιδευτικό σύστημα. Στο έγγραφο της Επιτροπή New Skills for New Jobs αυτό φαίνεται καθαρά. Και το ίδιο ισχύει και για τις ασκήσεις και μαθητείες. Πιο ενεργή πολιτική δηλαδή για την αγορά εργασίας τέλος οι επιχειρήσεις χρειάζονται επίσης κάποια στήριξη για τη χρηματοδότηση μαθητιών και ασκήσεων. Όσο για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, πολλές αγορές εργασίας είναι άκαμπτες. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μοιημένους να υποφεληθούν και αποκλείει τους καινούριου στην αγορά εργασίας και έτσι δεν γίνεται καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των νέων ταλέντων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε τώρα στα ερωτήματα των μελών. Πέντε είναι η πρώτη ομάδα. Η κυρία Λίν και μετά η κυρία Πασκαλούνια. Ε, εγώ φαντάζομαι ότι δεν μιλάμε για συγκεκριμένη έκθεση αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό έβαλα τον ε, λόγο μου εδώ πέρα για να αναφερθώ στην έκθεση, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι το οποίο εξέρχεται από τις παρεμβάσεις από την ETUC, από την ε, Business Europe, είναι να δώσουμε τις ε, δεξιότητες οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου εργασίας. Προφανώς η παιδεία δεν είναι θέμα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να μιλάμε για τους ασκούμενους και τους μαθητευόμενους, αλλά το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει προγράμματα τα οποία θα λειτουργήσουν στα κράτη-μέλη και πώς μπορούμε να μάθουμε κάτι από τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών. Όπως είπατε υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη, όπως φαίνεται και από την έκθεσή σας, από τα έγγραφα τα οποία μας έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια, όπου Λειτουργεί το σύστημα της μαθητείας, λειτουργεί το σύστημα των ασκουμένων πολύ καλύτερα από ό,τι σε άλλα κράτη-μέλη. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε αποκομίσει, γιατί δεν νομίζω ότι το κάνουμε αυτό με αρκετά επιτυχημένο τρόπο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο του να εξασφαλίσει ότι ό,τι είναι ήδη διαθέσιμο θα γίνει γνωστό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εξεταστεί από όλου για να δούμε και τα άλλα κράτη-μέλη που δεν έχουν αυτά τα συστήματα μαθητείας να τα εφαρμόσουν. Εγώ συμφωνώ να χρηματοδοτούνται θέσεις μαθητείας για θέσεις απασχόλησης οι οποίες έχουν μέλλον και όχι για αυτές που δεν έχουν μέλλον. Είναι σωστό αυτό. Και επίσης αυτά που έλεγχαν για τους ασκούμενους <clears throat> και εγώ πιστεύω ότι οι θέσεις ασκουμένων θα πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, παραδείγματος σε τρίμηνα, ότι θα πρέπει να είναι αμοιβόμενε οι θέσει αυτέ ασκουμένων, γιατί αλλιώ είναι μια μορφή εκμετάλλευση. Αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ξέρουμε τι γίνεται σε κάθε κράτο μέλο και δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει ένα μηχανισμό για να συγκρίνουμε τι πρακτικέ στα κάτι μελη Η κυρία Γκρουνή και η κυρία Μπλίνκεβιτ του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. για την έκθεση θα έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε συνεχεία. Θα συγκεντρωθώ λοιπόν στα ερωτήματα που έχω να θέσω προς τους ομιλητές και τους εμπειρογνώμονες. Τα παιδιά τα οποία έχουν αποτύχει στο σχολείο συνιστούν ένα πρόβλημα. Δεν θέλουν να συνεχίσουν το σχολείο. Τι μπορούμε να τους προτείνουμε. Γιατί συχνά είναι πολύ νέοι για να πάνε σε μια επιχείρηση. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να τους οδηγήσουμε σε μία λύση το συντομότερο δυνατόν. Τώρα για τον προσανατολισμό. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ιδέες τι είδους προσανατολισμό. Στη Γαλλία, επί παραδείγματι, ο προσανατολισμός ο δεν άλλαξε από τότε που εγώ ήμουν μαθητρία. Ε, θα επεξεργαστούμε κάποια κείμενα τώρα στη Γαλλία τώρα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε τον κόσμο του σχολείου με τον κόσμο της επιχείρησης. Ε, είναι δύο κόσμοι που δεν γνωρίζονται γενικά. Ε, τώρα με τις μαθητείες γνωρίζονται όλο και περισσότερο, αλλά γενικά παραμένουν χωριστοί κόσμοι. Έπειτα, η εξίσωση μεταξύ α, κατάρτισης και αγορά εργασίας. Ε, υπάρχει προσανατολισμός των νέων, τι θέλουν, να, τι θέλουν να κάνουν και τι μπορούν από τη μία και από την άλλη ε, τι απασχόληση θα τους προσφερθεί. Πίσω από όλα αυτά υπάρχουν τα νέα επαγγέλματα, αυτά που προτείνουμε σήμερα, αυτά που θα προτείνουμε σε 10 χρόνια, πώς μπορούμε να τα παντρέψουμε όλα αυτά και να δώσουμε στους νέους την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση. Έπειτα, ακούστηκε πολύ από κάποιους συναδέλφους ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσλαμβάνουν ε, μαθητευόμενους, θα, θα πρέπει να τους αμείβουν, θα πρέπει να τους διώχνουν. Ε, μια ερώτηση. Πώς θα τις βρούμε αυτές τις επιχειρήσεις. Εγώ έχω πάρα πολλούς νέους και γονείς που χτυπάνε στην πόρτα μου και μου λένε βοηθήστε με γιατί δεν ξέρω σε ποια επιχείρηση να στραφώ, σε ποια επιχείρηση να απευθυνθώ. Ευχαριστώ η κυρία Μπλίν και Βιτσούτε. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της και τους εμπειρογνώμονες και τους κοινωνικούς εταίρους για τις παρουσιάσεις τους. Συμφωνώ ότι είναι ουσιώδες το θέμα της ανεργίας των νέων να λυθεί και η Επιτροπή μας πρέπει να το διατηρήσει ως προτεραιότητα. Ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες της Ένωσης η ανεργία των νέων είναι υψηλότατη. Είναι τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα η ανεπιτυχής αρχή μιας καριέρα, επαγγελματικής καριέρας μπορεί να έχει τόσες αρνητικές ολόκληρη την ζωή του νέου και πρέπει ήδη από την αρχή της καριέρας αυτής να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος. Είναι σχεδόν αδύνατο αυτή τη στιγμή οι νέοι να μπουν στην αγορά εργασίας διότι το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν θέλει να τους απασχολήσει μόλις βγουν από το πανεπιστήμιο ή το γυμνάσιο εφόσον δεν έχουν εμπειρία. Το πρόβλημα λοιπόν για τους νέους, για την είσοδό τους δηλαδή στην αγορά εργασίας, είναι ότι είναι η μεταβατική περίοδος από την παιδεία, από την εκπαίδευση στην απασχόληση και αυτό μπορεί να είναι πολύπλοκο. Σε ευρωπαϊκό λοιπόν επίπεδο πρέπει να ληφθούν νέες πρωτοβουλίες ώστε να μάθουν οι νέοι την κινητικότητα και να ακολουθήσουν κατάλληλες ασκήσεις και μαθητείες. Σε εθνικό δε επίπεδο το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να βελτιωθεί διότι οι δεξιότητες και η κατάργηση πρέπει να ακολουθούν και τις δυναμικά αλλά αλλάζουσες συνθήκες της αγοράς εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Χίρς και μετά η κυρία Φιγκερέιντο. Εσείς, κυρία μου, που μιλήσατε και πριν, τελευταία. Η κυρία Χίρς, δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ χρήσιμο το ότι ζητάμε συζητάμε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο γίνεται στις χώρες μας όλο και πιο επίκαιρο. Αλλά φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει από εξανέκαθεν, δεν είναι καινούριο. Θα πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ των νέων, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο αποχωρούν πρόωρα από το σχολικό σύστημα, γιατί το σχολικό σύστημα δεν είναι κατάλληλο για αυτούς. Έχουμε το πρόβλημα αυτό της πρόωρης αποχώρησης. Αυτό ίσως είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν προέρχεται από τους ε, ίδιους τους νέους. Είναι απαραίτητο να δώσουμε μεγαλύτερη δημιουργικότητα στο σχολείο και να δώσουμε στους νέους την ενθάρρυνση να χρησιμοποιήσουν τις πραγματικές τους ικανότητες στο σχολείο και να κάνουν κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει κιόλα. Ότι πρέπει να επενδύσουμε στην κατάρτιση. Αυτό το ακούω από τότε που είμαι πολιτικά ενεργή, αλλά στην πράξη ποτέ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε προγράμματα υποδείγματα ένα, δύο, τρία χρόνια έχουν αυτή την επιτυχία, αλλά μετά δεν υπάρχει καμία συνέχεια η οποία πρέπει να δοθεί. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι με επιτυχία τελειώνουν αυτά τα προγράμματα δεν τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν καλές θέσεις εργασίας. Από την άλλη πλευρά είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μια καλή παιδεία και έχουν απλώς μια ακαδημαϊκή κατάρτιση αλλά δεν έχουν καμία απολύτως πρακτική πείρα. Πρέπει λοιπόν γι' αυτό το λόγο να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των δύο αυτών καταστάσεων. Θα πρέπει εδώ να ξέρω από την πλευρά των ε, εμπειρογνωμόνων πόσο μπορεί να υπάρξει πρόβλημα παραγωγός χάρη με την ε, νομοθεσία η οποία πολλές φορές δεν επιτρέπει στους νέους να εργάζονται. Να είναι ας πούμε εργαζόμενοι μόνο σε ένα περιορισμένο επίπεδο γιατί λένε πολλές φορές οι εργοδότες 16 χρονών είναι πολύ νέος κανείς για να εργαστεί θα πρέπει να κάνει μια μαθητεία και να επανέλθει αργότερα παραγωγικά στην ηλικία των 18. Δηλαδή πολλές φορές φοβάμαι ότι οι ρυθμίσεις οι οποίες υπάρχουν νομοθετικά στις χώρες μας μπορεί να εμποδίσουν και την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Κύριε Φιγκυρέντου. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ σημαντική είναι αυτή η συζήτηση, γιατί σήμερα η ανεργία των νέων είναι μια μεγάλη ανησυχία για όλους μας. Πάνω από 21% των νέων μας είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή. Και συμφωνώ με αυτά τα οποία ελέγχθησαν από πολλούς, ότι τα στάζ δεν πρέπει να είναι φτηνή παροχή εργαζομένων στις επιχειρήσεις και το καθεστώς αυτών οι οποίοι είναι στη, στα προγράμματα άσκησης μαθητείας θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα. Να υπάρχει λοιπόν ένα χρονικό πλαίσιο, να υπάρχει μια αμοιβή των ασκουμένων, ώστε να μην συνεχίσουν οι επιχειρήσεις να αντικαθιστούν τους εργαζομένους τους από ασκουμένους που τους αλλάζουν κάθε τόσο, όπως φάνηκε να γίνεται πολλές φορές στην Πορτογαλία. Θα ήθελα εδώ να έχω τα σχόλιά σας. Δεύτερο θέμα είναι αυτό που έχει να κάνει με την επαγγελματική κατάρτιση και κυρίως με το θέμα του πώς αντιμετωπίζουμε τη σχολική αποτυχία. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι είναι πολλοί οι παράγοντες που οδηγούν στην σχολική αποτυχία. Πολλές φορές η ίδια η παιδεία δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των νέων, τους στόχους τους και όλα αυτά. και πολλές φορές η λειτουργία των σχολείων αντανακλά τα κοινωνικά προβλήματα, την ανεργία, την ένδια κτλ. Δεν μπορούμε λοιπόν να απομονώσουμε το θέμα της σχολικής αποτυχίας και της εγκατάλειψης της πρόορης των σχολείων από τον περίγυρο των κοινωνικών προβλημάτων που υπάρχουν σε μια κοινωνία. Θα πρέπει να δούμε γιατί υπάρχει υψηλό επίπεδο σχολικής αποτυχίας σε ορισμένες περιπτώσεις και να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του κακού, όχι να πούμε ότι θα πρέπει κάποιος ο οποίος δεν πάει καλά στο σχολείο να κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν ένας μεγάλος αριθμός λύσεων που ακόμα και το σχολείο μπορεί να δώσει και ξέρω πολλές περιπτώσεις που έχουν υπάρξει θετικές λύσεις. Μερικά από αυτά τα προγράμματα έχουν πετύχει, αλλά όχι. Ευχαριστώ, θα σας δώσω και πάλι το λόγο. Ζητών από εσά να απαντήσετε σε βαθμό, σε πιο συνοπτικό τρόπο. Πρέπει να πω να απαγορευτούν οι θέσεις άσκησης εάν δεν δίνουν επαγγελματικά προσόντα, εάν δεν δίνουν διπλώματα. Τι πιστεύετε σε σχέση με τις προτάσεις της κυρίας Τουρουνέν που λέει στην αιτιολογική της σκέψη ΤΑΦ, ότι πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο αποδοχών για τους νέους, ότι μάλλον το ελάχιστο αυτό επίδομα το οποίο δίνεται στους νέους στη Δανία, Ενωμένο Βασίλειο και Γαλλία, τους εμποδίζει να μπουν στην αγορά εργασία. Βέβαια τα κακά νέα είναι ότι έχετε μονάχα δύο λεπτά για να απαντήσετε ο καθένα σας. Γιατί αν δώσω το λόγο στους νέους μετά, τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση, τι νόημα έχει αυτή η συνάντηση. Δύο λεπτά. Έχω πολύ ωραία τέσσερα σημεία για να αντιδράσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, για τις μαθητείες και το στάζ. Δεν επανέρχομαι στην, στον ορισμό του καθηγητή ΜΕΝΚ, συμφωνώ. Ε, βεβαίως θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε την ε, μαθητεία από την άσκηση. Για, το, για τη μαθητεία. Θέλω να τονίσω το εξή ότι το, η μαθητεία θα πρέπει να πλαισιώνεται, να υπάρχει μια σύμβαση, να πληρώνεται και δεν θα πρέπει ε, να υποκαθιστά ε, μια πραγματική θέση απασχόλησης. Δεν θέλουμε δηλαδή φτηνούς ε, εργαζόμενους ε, παύλα μαθητευόμενους. Έπειτα, για να υπάρχει ωστόσο προσανατολισμός πρέπει να υπάρχει επιλογή. Για να ε, επιλέξει μια επαγγελματική σταδιοδρομή ένας νέος θα πρέπει να ξέρει τον περιμένει. ενημέρωση λοιπόν για τις διεξόδους, αν ασχοληθώ με την ψυχολογία ή με, γίνω μηχανικός, τι λύσεις υπάρχουν στο τέλος, τι δουλειά μπορώ να χτυπήσω στο τέλος. Ε, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να κάνουμε τους νέους πρόβατα, ας πούμε, αλλά να τους να δώσουμε τη δυνατότητα να επιλέξουν. Εγκατάλειψη του σχολείου τώρα. Θέλω να μιλήσω για κάτι περίπλοκο, ε, το οποίο αναφέρθηκε, το πλαίσιο της οικονομικής ε, κρίσης, που θέτει τους νέους σε δυσκολία. Οι δυσκολίες αυτές που αντιμετωπίζουν οι νέοι έχουν να κάνουν με τη συγκυρία, με τις δυσκολίες στην αγορά απασχόλησης. Ε, γι' αυτό θέλουμε να υπάρχουν ε, πολιτικές ε, στο χώρο της αγοράς εργασίας, ενσωματωμένες, ολοκληρωμένες. Τέταρτο σημείο. Ε, νομοθεσία για την απασχόληση των νέων. Ε, θα υπομοιδιάσω λιγάκι για αυτό το σημείο. και η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Σήμερα όταν βλέπουμε το επίπεδο ανασφάλεια των νέων και επισφαλών θέσεων ε, απασχόληση. Αυτό που θέλουμε για τους νέους τι είναι. Πλαισίωση, ε, ασφάλεια και, και διαπραγματεύσεις για τους νέους. Αυτό είναι ο βασικός κανόνας. Έτσι. Να εξασφαλίσουμε μια ασφαλή θέση απασχόλησης. Ε, τέσσερις απαντήσεις, ε, τέσσερις διαδρομές σε δύο λεπτά. Μπράβο. Ο επόμενος μπορεί να μιλήσει εξίσου γρήγορα να αρθεί στο ύψος της πρόκλησης. Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω. Πρώτον, το σύνολο της εκπαίδευσης ενός νέου, η διαβίου μάθηση και τα λοιπά, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε έτσι σφαιρικά. Γιατί είναι πιο πολύπλοκο από απλή εκπαίδευση στην αρχή της ζωής. Το θέμα είναι στους νέους από την νεαρότερη δυνατή ηλικία της συνείδησης ότι πρέπει να συνεχίσουν να μετεκπαιδεύονται γιατί στην αγορά εργασίας αλλάζουν ραγδαία τα πράγματα και πρέπει και εκείνοι να αλλάζουν. Το θέμα λοιπόν είναι η συνειδητοποίηση του γεγονότος αυτού από τους νέους τη στιγμή, από τη στιγμή που μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Άλλο θέμα. Είναι όλο και μεγαλύτερη η σημασία που δίνεται στα λεγόμενα soft skills. Πολλοί δεν το δέχονται αυτό. Γιατί η παραγωγικότητα της εργασίας, οι σχέσεις τους, οι πελατειακές τους σχέσεις και τα λοιπά είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει ανάλογα με τα γενικά αυτά soft skills. Τώρα για την πραγματική είσοδο στην αγορά εργασίας, οι μαθητείες και οι ασκήσεις. Στην πραγματικότητα είναι διαφορετική η κατάσταση που ισχύει για αυτά από χώρα σε χώρα. Και η συζήτηση του θέματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι μπορεί να δείξει. Μπορούν να ταυτιστούν μερικά προβλήματα ή ελλείψεις, αλλά σχετικά με το τι δουλεύει πράγματι στην πράξη, αυτό, αυτό σχετίζεται με τη δυνατότητα ενός ασκούμενου να έχει πραγματικά εργασιακή εμπειρία, όχι θεωρητική κατάρτιση. Αυτό το καταλαβαίνουν οι νέοι ότι αυτά που πρέπει να μάθουν είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσουν πράγματι στη δουλειά τους αργότερα. Α, έλξε ο χρόνος είναι να σας κάνω. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε στο τρίτο τμήμα αυτής της μακροσκελούς ακρόασης το πιο δύσκολο ίσως γιατί επειδή χρειάζεται αυτοπιθαρχία σε όλους επειδή υπάρχουν πολύ προσκεκλημένοι από το γραφείο, από το φόρουμ μάλλον των νέων Ευρωπαίων δίνω το λόγο στον κύριο Λουκά Καρπιέλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τουρούνεν που μας προσεκάλεσε σε αυτή τη συζήτηση για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση της κρίσης, η οποία δημιουργεί μεγάλα προβλήματα για όλους τους νέους στην Ευρώπη. Και σαν οργάνωση νέων έχουμε να κάνουμε πολλά και να πούμε πολλά σχετικά. Συμφωνούμε όλοι ότι η κρίση θέτει ένα αμφιβόλο την κατάσταση των νέων ανθρώπων. Και οι νέοι είναι μια από τις πιο τρωτές ομάδες στην κοινωνία και εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον έγγραφο της Κομισιόν που λέει για την κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη που λέει σαφώς ότι είναι οι νέοι οι οποίοι πλήττονται περισσότερο. Τώρα έχουμε 21,4% ανεργία ενώ έχουμε ξεκινήσει από 16,4% πριν από 6 μήνες. Αυτό δείχνει ότι πράγματι υπάρχει κάτι το οποίο αρχίζει να ραγίζει μέσα στον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης ό,τι αφορά τους νέους και πρέπει να το σκεφτούμε αυτό τώρα που συζητούμε για το ποια θα πρέπει να είναι η νέα οικονομική στρατηγική, στρατηγική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης πιστεύω ότι εφόσον μιλάμε εμείς για τα θέματα της μετάβασης, του επιχειρήν, της ε, θέσης εργασίας με ποιότητα, πρέπει και αυτά τα στοιχεία να προσθεθούν στη συζήτηση και όχι να παραμείνουμε στα πλαίσια αυτών που τα γνωρίζουμε. Είναι απαραίτητα αυτά ιδίως σε καιρούς κρίσης. Θέλω να απαντήσω σε σχέση με ορισμένα σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μένα. Για τις θέσεις άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Νέων ασχολείται με τα θέματα αυτά από το 2008. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αποφύγουμε αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Οι θέσεις ασκουμένων, ιδίω πέραν και έξω από το σύστημα εκπαίδευσης, αντικαθιστούν τις αμοιβόμενες θέσεις εργασίας γιατί ιδίω σε χώρε όπω η Ιταλία και η Γαλλία οι επιχειρήσει αντικαθιστούν του αμοιβόμενου εργαζόμενου με του ασκούμένου. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε γιατί δεν είναι αυτό το νόημα που έχει μια τέτοια θέση άσκηση. Η άσκηση πρέπει να είναι μια ευκαιρία, ένας χρόνος παιδεία και άσκηση με μια εταιρεία ατόμων με πολύ ισχυρό και προχωρημένο επαγγελματικό προφίλ που αποκομίζουν περισσότερες δεξιότητες. Σε καιρό κρίσης δεν είναι χρήσιμες οι θέσεις ασκουμένων για το σκοπό αυτό. Και τώρα πρέπει να περάσουμε από τις δεσμεύσεις μας στις δράσεις. Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε μια δέσμευση να σκεφτεί και να προβληματιστεί για το θέμα αυτό. Τίποτα δεν έχει προέλθει όμως μέχρι στιγμής. Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος για τους νέους 2020 θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νέων προτείνει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για ένα νέο πλαίσιο για τις θέσεις άσκησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν δύο κύρια είδη άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι οποίοι ασκούνται μέσα στον εκπαιδευτικό τομέα και οι άλλοι που ασκούνται εκτός του εκπαιδευτικού τομέα. Μπορεί να είναι διαφορετικοί στόχοι, αλλά είναι ίδιες οι ανάγκες των ασκουμένων και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με ευελιξία. Ένα άλλο σημείο που για μένα είναι πολύ σημαντικό, αυτό που έλεγε η Business Europe, είναι το θέμα των υπείων δεξιοτήτων, των soft skills. Δεν είναι αυτά τα πράγματα που μαθαίνει κανείς μόνο με την τυπική παιδεία. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα σύνορα της τυπικής με την ατυπική παιδεία. Είναι απαραίτητο να επενδύσουμε στο τι μπορεί να επιτύχει κανείς από άτυπα εκπαιδευτικά κανάλια οι δεξιότητε που μπορεί να αποκομίσει κανεί παγκοσχάρη εργαζόμενο για μια μη κυβερνητική οργάνωση. Επομένω, χρειάζεται μια καλύτερη επαλήθευση των προσόντων των νέων. Και υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία τα οποία είναι για μένα σημαντικά. Καταρχήν η συζήτηση για το πώ να εξασφαλίσουμε καλύτερε απαντήσει των νέων για τα προβλήματα κοινωνική προστασία και την πρόκληση τη ευέλικτη Τι θα κάνουμε λοιπόν μεταξύ μιας εργασίας βραχίας διαρκείας και μιας άλλης εργασίας βραχίας διαρκείας. Γιατί τώρα ακόμα και δεν υπάρχει ιδιαίτερη επένδυση από τα κράτη-μέλη για να καλυφθεί αυτό το χάσμα, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και επίσης υπάρχει το άλλο πρόβλημα το οποίο αναδείται στην Ευρώπη, ότι φεύγουν οι νέοι από τον οικογενειακό χώρο αργότερα, χάνουν την αυτονομία τους είναι σε κίνδυνο η αυτονομία των νέων στην Ευρώπη. Και ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι να χρησιμοποιήσουμε υποφελέστερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Γιατί αυτό είναι το καλύτερο εργαλείο που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως είναι η ανεργία και να έχουμε θέσεις ασκουμένων με ποιότητα και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτών που φεύγουν πρόωρα από το σχολείο. Πρέπει να έχει καλύτερη στοχοθεσία σε σχέση με τους νέους τους οποίους αντιμετωπίζει και αυτή η συζήτηση θα πρέπει να είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει μέσα στα πλαίσια της νεότητος 2020 και να είναι ένα στιγμίο προβληματισμού. Θέλω να σταματήσω εδώ γιατί έχω ξεπεράσει το χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ για το Generation Précaire αβέβαιη γενιά, ο κύριος Γιάννικ Μιέλα. Πέντε λεφτά. Είναι ενδιαφέρον να συζητάμε για τους νέους όπως σήμερα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ε, από τη μία καλή θέληση από τους πολιτικούς, έτσι τουλάχιστον ε, ισχυρίζονται, και από την άλλη όμως η πραγματικότητα των νέων είναι τελείως διαφορετική. Ε, Παρ' όλα αυτά πρέπει να επενδύσουν στο μέλλον των νέων. Στο μέλλον των νέων. Είναι οι μελλοντικοί εργαζόμενοι. Αλλά στη Γαλλία έχουμε ένα, μια περιφρόνηση ψυχολογική και περιφρόνηση από τον νόμο. Ε, έχουμε τους νέους της γενιάς Y ε, σε ένα από τα γαλλικά site ε, γράφανε, γράφανε διάφορα σχόλια ότι, για μας, αυτή τη γενιά, ότι έχουν κίνητρα, αλλά το κίνητρο τους είναι βασικά το χρήμα, είναι βιαστική, είναι αδιφάγη κτλ. Αυτά λένε για μας. Το δεύτερο είναι ο νόμος. Στη Γαλλία υπάρχει κάτι που προβλέπεται από τον νόμο, ένα συμπλήρωμα δηλαδή, ε, για να συμπληρώσει το, κανείς το εισόδημά του. Αλλά πρέπει να είναι 25 ετών τουλάχιστον για να του δοθεί αυτό το συμπλήρωμα. Δηλαδή, όχι πολύ νέος τελικά. Ε, ε επίσης, ο αριθμός των σταζιέχ, των μαθητευόμενων, ε, είναι πέρασε από τους 800.000 στο 1,2 εκατομμύρια. Ε, επίσης ο νόμος λέει ότι δεν καλύπτονται από τον εργατικό νόμο. Επίσης, ε, αν το στάζ διαρκεί πάνω από δύο μήνες, είναι 400 ευρώ. Ε, είναι κάτω από το 50% του κατοφλίου φτώχειας ο μισθός που παίρνουν, η απολαβή τέλος πάντων που παίρνουν οι ε, σταζιέ. Έχουμε 1,2 σταζιέ στις επιχειρήσεις, εκατομμύρια στις επιχειρήσεις. Ε, η Γαλλία βεβαίως ξέρουμε ότι είναι υπερχρεωμένη ε, και δεν συνεισφέρει το κράτος για τις συντάξεις αυτών των νέων. αυτοί οι νέοι ούτως ή άλλως δεν έχουν χρήματα για να καταναλώσουν, τρέχονται άσχημα και οι ίδιοι επίσης δεν συνεισφέρουν για τις μελλοντικέ τους συντάξεις. Επομένω, ούτε το κράτος βοηθάει τους νέους, ούτε οι νέοι τον εαυτό του. Επίσης έχουμε ένα άλλο καλό σύστημα, την άσκηση, που λειτουργεί στη Γαλλία θαυμάσια. Ιστορικά είναι πλαισιωμένο αυτό το, το σύστημα. Η Έμιλη Τουρούνεν έχει μια θαυμάσια ιδέα. Ε, ανάφερε στην ίδια έκθεση τις μαθητείες και τις ασκήσεις. στη Γαλλία δεν μπορούμε να τα δούμε και τα δύο συστήματα παράλληλα το, τα βλέπουμε τελείως χωριστά, αποκομμένα. Χρηματοδοτούμε άνετα, έτσι γενναιόδωρα την άσκηση, αλλά αγνοούμε και υποχρηματοδοτούμε τη μαθητεία. Ένας μαθητευόμενος ε, δεν κοστίζει τίποτα σε, σχέση με έναν ασκούμενο. Ένας στα κοστίζει έξι φορές λιγότερο από τον εργαζόμενο, αλλά κοστίζει και λιγότερο και από τον ασκούμενο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την ανάπτυξη της άσκησης χωρίς να μιλήσουμε για την πλαισίωση της στάζ. Εγώ δεν θέλω να συνεχιστεί αυτό το στάζ όπως υπάρχει στη Γαλλία. Δεν μπορούμε να βάζουμε τους νέους σε επιχειρήσεις και να λέμε ότι δεν καλύπτωται από το εργατικό δίκαιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λέμε ότι το, το στάζ είναι μια περίοδος μαθητείας, ε, άσκησης απ' την άλλη. Α, έτσι το ορίζουμε. Πηγαίνετε στο ίντερνετ, κοιτάξτε τις προσφορές για την ε, μαθητεία ε, και για να κάνει κανείς... Ε, έχει κανείς μια τέτοια περίοδο μαθητείας, βασικά πρέπει να είναι διπλωματούχος, να έχει πάρει το πανεπιστήμιο, όσο κακό και να είναι, και να έχει και εμπειρία για να κάνει στάζ παρακαλώ. Επομένως, πρέπει να κάνουμε κάποια χειρονομία. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο μισθό για το σταζιέρ ε, σε σχέση με τον ελάχιστο μισθό των εργαζομένων. Δεν μπορούμε να του ε, αποδγυμνώσουμε, αποδυναμώσουμε από την ελάχιστη εργατική προστασία. Ε, επαναλαμβάνω, 1,2 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται στις επιχειρήσεις και δουλεύουν στα ΣΓΕ ε, με πάρα πολύ άσχημους όρους. Οι επιχειρήσεις ε, λένε, φανταστείτε αν πληρώνουμε 1,2 εκατομμύρια άτομα, ε, υπάρχει πρόβλημα. το θέμα είναι να βάλουμε τους σταζιέρ σε θέσεις απασχόλησης με προοπτική, αλλιώς να μην υπάρχει στάζ. Εγώ νομίζω ότι το σημερινό στάζ με τη σημερινή του μορφή είναι μια, φωτή, μια μορφή δουλειά. να καταργηθεί. Σας ευχαριστώ για τα λόγια αυτά που είπατε έξω από τα δόντια. Θα σας προτείνω την εξή μέθοδο. Τα επόμενα δύο άτομα θα μιλήσουν, αυτά που μου ζήτησαν το λόγο δηλαδή, πρώτοι, και συνέχεια θα κάνουμε ένα μικρό γύρο τραπέζις, ούτως ώστε κάθε ομάδα να μιλάει ε, και να τοποθετηθεί πάνω στην έκθεση του Ρούνεν. Και η κυρία του Ρούνεν θα παίρνει τελευταία το λόγο για να κλείνει τη συζήτηση, έτσι, τμηματικά. Πολύ ωραία, αν συμφωνείτε. Συμφωνείτε. Ε, ο κύριος Κρίστανσεν και μετά η κυρία Ντελή. Α, όχι τότε η κυρία Ντελή κατευθείαν. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με την οργάνωση Generation Precaire πρέπει να υπάρξει κάποια πλαισίωση των μαθητιών και ασκήσεων. Γιατί νομίζω ότι η νεολαία ζει έναν μόνιμο αγώνα στον οποίο είναι χαμένη από χέρι. Δεν έχει κοινωνικό καθεστώς αναγνωρισμένο, ούτε, ως ούτε οι φοιτητέ το έχουν κάνει. Και όταν μπαίνουν στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζουν τρομερές συνθήκες. Να σας πω ποιες είναι. Οι νέοι που μπαίνουν στην αγορά εργασίας λοιπόν έχουν χαμηλούς μισθούς για ίσες δεξιότητες, δεν έχουν μόνιμο καθεστώς και ιδίω έχουν συνθήκες εργασίας χειρότερες από τους άλλους. Και οι απαιτήσει του εργοδότη είναι συνήθως τελείως παράλογες έγινε λόγος για το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Ανέχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Ε, αυτό το θέμα η Επιτροπή μας νομίζω ότι πρέπει να το στηρίξει και να αρχίσει να το συζητάει συγκεκριμένα. Το εισόδημα αλληλεγγύης, όχι σύμφωνα με το γαλλικό σύστημα, αλλά ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για όλους, γιατί είναι απαράδεκτο σήμερα να, όταν κανείς γίνεται 18 ετών να χρειάζεται να περιμένει χρόνια ολόκληρα για μέχρι να βρει κάποια ευημερία να πετύχει σε εισαγωγικά διότι οι νέοι είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης και για τη στέγαση αναγκάζονται να καταλήγουν σε ειδικέ κατοικίες για τους πτωχότερους και η διαδικασία της Βολονίας ίσως να βοηθούσε γιατί η ανέχεια τους αφορά όλους, όλους. Και αυτό πολύ σημαντικό, και αυτό. Και αυτό. Διότι η διαδικασία της Βολονίας είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει το υπάρχον και ανεπαρκές εκπαιδευτικό σύστημα. Ευχαριστώ. Τώρα θα γίνει ο γύρος των ομάδων. Παρακαλώ να μιλήσετε και σε απάντηση όσων είπαν οι δύο εκπρόσωποι των οργανώσεων και, και για την έκθεση του Ρούνεν καθεαυτήν, Νταζάιν έκθεση του Ρούνεν. Λοιπόν, δύο λεπτά ο καθένας για το ΕΛΚ. Ε, η κυρία Γκρουνή, πως η κυρία Φοντανιέ, ποια από τις δύο, ποια από τις δύο. Τις δύο για την ε, έκθεση αυτή λοιπόν της κυρίας Τουρούνεν. Ε, προφανώς θέλω να την ευχαριστήσω και να τη συγχαρώ για την ποιότητα της εργασίας της. Νομίζω πρέπει να επιμείνω στο σημείο της προσαρμογής, της κατάρτισης, της ανάγκης της αγοράς, όπου αναφέρθηκε και προηγουμένως. Για τα στάζ, εγώ έχω ακούσει πάρα πολλά σήμερα τα στάζ είναι σημαντικά σαν πρώτη παροχή εμπειρίας για τους νέους, αλλά είναι μια πρώτη εμπειρία μονάχα. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια διάκριση μεταξύ αυτών και της μαθητείες που δίνουν ένα δίπλωμα στο τέλος, τα στάζ δεν το κάνουν αυτό. Η αμοιβή στα στάζ, θα σας έλεγα να μην το ενσωματώσουμε αυτό στη συζήτηση, γιατί δεν ξέρω αν θα πρέπει να έχουμε αμοιβόμενους σταζιέρ σε μια επιχείρηση ή μη αμοιβόμενου. Για μένα το ουσιαστικό είναι ότι όταν τα στάζ αυτά γίνονται σε ένα επίπεδο χάρη τρίμηνο, προσφέρουν κάτι σε μια επιχείρηση και τότε θα πρέπει να υπάρχει κάποια αμοιβή η οποία εξαρτάται από το είδος του στάζ. Λιγότερο από τρεις μήνες εκεί πράγματι περισσότερο δίνει η επιχείρηση στον σταζιέρ, χρειάζεται χρόνος από την επιχείρηση για να δώσει τις γνώσεις των ασκούμενο στο στάζ και τότε νομίζω ότι δεν είναι η επιχείρηση η οποία πρέπει να πληρώνει, μάλλον πρέπει να πληρώνεται. Ε, πρέπει να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ ΣΤΑΖ και επιχείρησης. Γιατί θα ήταν προς ζημία των νέων να μην βρίσκουν μια επιχείρηση για να κάνουν στάζ. Εγώ νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτή η προσέγγιση μεταξύ νέων και επιχειρήσεων. Επίσης, για την έκθεση της κυρίας Τυρινέν, πέραν του θέματος της αμοιβή ή όχι, μια μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε με τους νέους όταν είναι στα πλαίσια ενός στάζ, βρίσκεται το θέμα της κινητικότητα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει και μια βοήθεια αυτοί οι νέοι που είναι σε στάζ για να μπορέσουν να μετακινηθούν και να έχουν στέγαση στον τόπο εργασίας τους. Πιο σημαντικό είναι αυτό από την αμοιβή. Γιατί πολλέ φορέ δεν έχουν την δυνατότητα να πάνε στον τόπο αυτό που θα του δώσει την καλύτερη πρόσβαση στι επιχειρήσει που έχουν να του προσφέρουν κάτι. Και εδώ ίσω θα ήταν πολύ σημαντικό να του βοηθήσουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Αυτά ήθελα να πω. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση η οποία καταλαμβάνει πολλά στοιχεία σημαντικά και σίγουρα θα προωθήσει τα πράγματα. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες τώρα. Ο Σύντομα, Πρόεδρε. Ε, έχουμε υποβάλει και προπολογίες. Η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μας άνοιξε πολλούς δρόμους προβληματισμού. Ε, δύο πράγματα θέλω να τονίσω ε, στην εισηγητριά μας. Καταρχάς, μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μετάφρασης στο εκτιμώντας F σιγματάφ τότε πρέπει να το αλλάξει. Γιατί εγώ δεν νομίζω ότι το ελάχιστο εισόδημα ένταξης είναι αυτό που εξασφαλίζει μία ανεξάρτητη ζωή στον νέο. Όχι. Δεν νομίζω ότι τα επιδόματα του εξασφαλίζουν ανεξαρτησία, εξαρτησία. Αν δεν μπορεί ας πούμε, το οικονομικό σύστημα να τον εξασφαλίσει, προσοχή ε, στα επιχειρήματά μας, έτσι γιατί παρότι έχουμε καλή θέληση, δεν πρέπει να κλείνουμε το, και να στρέφουμε την πλάτη μας στις λίγες ευκαιρίες που έχουν οι νέοι για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω του οικονομικού συστήματος. Αυτά που είπαν οι νέοι εκπρόσωποι ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπω ότι η συγγήτρια που είναι Δανέζα είναι πολύ ικανοποιημένη από το πώς ε, λειτουργεί η, η ασφάλεια και η ευελιξά ασφάλεια στη Δανία. Ε, πρέπει να τα δούμε όλα μαζί. Ε, το κοινωνικό σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα. Γιατί αλλιώς οι νέοι θα έχουν πραγματικά λίγη ασφάλεια. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Η λίγη ασφάλεια. Και όχι πολύ ευέλικτη ασφάλεια. Και τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε μια Ευρώπη προοδευτική που δημιουργεί απασχόληση, δραστηριότητα για τους νόους, ένα καλό πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων, προς κοινωνικής προστασίας, πέρα από τις ειδικέ πολιτικές για τους νέους. Έτσι. Χρειαζόμαστε αυτή την Ευρώπη. Ευχαριστώ για τους φιλελεύθερους. Η κυρία Χίρσ. Και εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε για αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι έχει πολύ καλές προτάσεις. Μία από τις δυσκολίες είναι ότι πάλι πρέπει να εξαρτιόμαστε από τη δράση των κρατών μελών. Είναι περιορισμένη η δυνατότητά μας παρέμβαση λόγω της επικουρικότητας και αυτό είναι κρίμα. Αυτό όμως που πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά είναι η χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Υπάρχουν πολλά σε διάφορα μέρη προγράμματα και σχέδια τα οποία λειτουργούν και ίσως θα πρέπει εδώ να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη σύνδεση αυτών των σχεδίων με την απασχόληση των νέων. Σε ό,τι αφορά τις μαθητείες και την άσκηση μάλλον, αυτό θα πρέπει να το διαχωρίσουμε από την ε, εκπαίδευση εν κενό αέρος κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να δούμε την ε, άσκηση σαν τμήμα της ε, εκπαίδευσης. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι τμήμα της εκπαίδευσης και κάποιος ο οποίος ασκεί θα πρέπει να μάθει κάτι μέσα σε αυτό. Όταν έχει μεγαλύτερη διάρκεια από ένα όριο, αυτό πια δεν είναι άσκηση, είναι μια μορφή εργασίας και παροχής εργασίας. Και επομένως αντικαθιστά θέση εργασίας σε μια επιχείρηση. Τώρα, το κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε είναι ότι η ανεργία οδηγεί και σε προβλήματα, σε άλλα προβλήματα για τους νέους σε σχέση με το εισόδημα το οποίο προσδοκούν στη συνέχεια αυτοί που είναι μακροχρόνια άνεργοι παραγωγός χάρη, μειώνουν κατά ανάγκη τους, ε, τις ε, προσδοκίες τους και εν καιρό δεν θα έχουν και επαρκείς ε, συντάξεις γιατί δεν θα έχουν συν, δεν θα έχουν μαζέψει τις ώρε εργασία που είναι απαραίτητες. Και εξάλλου αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μια αρνητική επίπτωση στο βιογραφικό ενό νέου, το να έχει μείνει άνεργος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλω και πάλι λοιπόν να συγχαρώ την εισηγήτρια. Merci. Σας ευχαριστώ. Κυρία Τουρούνε, θα σα δώσω το λόγο στο τέλος, έτσι. Από την ΚΟΕ, κυρία Φιγκερέιδο. Δεν είναι υποχρεωτικό, ε. Μου αν θέλετε. Δύο πράγματα πάρα πολύ σύντομα θέλω να πω. Γιατί έχουμε καθυστερήσει. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση υπήρξε εξόχω σημαντική και ενδιαφέρουσα γιατί μα έφεραν οι νέοι τι δικέ του εμπειρίε και τι ζωντανέ πτυχέ τη πραγματικότητα που ζουν. Και εμεί πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη στην έκθεσή μα υπό τη μία ή την άλλη πτυχή του θέματος. Χρειάζεται λοιπόν η έκθεση να προσαρμοστεί και να λάβει υπόψη τις εμπειρίες που μας ανέφεραν οι νέοι. Ελπίζω θα μας αφήσουν και έγγραφες μορφές των παρεμβάσεών τους για να μπορέσουμε να τις λάβουμε υπόψη μας κατά τη συζήτηση της έκθεσης της κυρίας Τουρούνεν. Η κυρία Τουρούνεν. Ευχαριστώ. Όλους τους συναδέλφους και τους προσκεκλημένους μας. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που ήρθατε εδώ και που βοηθήσατε στην έκθεση. Ευχαριστώ και την ε, γραμματεία. Ήταν πολύ ευέλικτη και στη διάθεσή μας. Και ε, το πιο σημαντικό από όλα ήταν ότι συμμετείχαν και εκπρόσωποι των νέων. Ε, είναι σημαντικό να συμμετέχουν εκπρόσωποι των νέων κάθε φορά που συζητάμε τις πολιτικές για τους νέους. Τώρα, οι σοσιαλιστές θα πρέπει να διαβάσουν πιο προσεκτικά την έκθεση, γιατί αυτό που είπα για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία και τη Γαλλία είναι ότι αν υπάρχει ειδική νομοθεσία για τους νέους, ειδική, που δεν τους επιτρέπει να δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη και ενήλικη ζωή, υπάρχει πρόβλημα το ελάχιστο εισόδημα για τους νέους ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο κάτω των 25 είναι πολύ χαμηλό. Δεν μπορούν να ζήσουν πραγματικά αξιοπρεπώς με αυτό. Απλώς τα τονίζω αυτά τα προβλήματα, τα υπογραμμίζω. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ξανά το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί θέτει ψηλά στις προτεραιότητές του το θέμα της ε, δημιουργίας τη απασχόλησης. Τώρα για την ευέλικτη ασφάλεια. Τι είπα? Ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτή την τραγωδία Ε, υπάρχει ανισορροπία ανάμεσα στην ε, ευελιξία και στην ασφάλεια. Το ξέρουμε, συμφωνούμε. Και η μετάβαση προς την ασφάλεια πρέπει να είναι η λέξη κλειδί. Μετάβαση προς την ασφάλεια. Ε, θα πρέπει απλώς να διορθώσουμε τα πράγματα. Επίσης, στην έκθεση πρέπει να τονίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στην μαθητεία και την άσκηση και θα κάνω και εγώ δικές μου τροπολογίες στην έκθεσή μου για αυτό το σημείο γιατί είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας σχόλια. Νομίζω ότι μπορώ να τα εντάξω σε μεγάλο βαθμό στην έκθεση χωρίς πρόβλημα. Και τέλος κάτι περίπλοκο. Ξέρω ότι δεν έχουμε αρμοδιότητες ε, για την εκπαίδευση. Η νεότητα είναι ένα οριζόντιο πρόβλημα. Ε, μιλάμε για την εκπαιδευτική πολιτική, α, τις μακροοικονομικές πολιτικές, κοινωνικές πολιτικές, πολιτικές για την απασχόληση και όλες αυτές θα πρέπει να τις συγκεράσουμε σε πολιτικό επίπεδο. Και αυτή είναι η βασική πρόκληση. Σε αυτή την Επιτροπή θα πρέπει, και εδώ αναλαμβάνω τις δικές μου τις ευθύνες ως συγκήτρια, θα πρέπει να δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι μπορούμε να κάνουμε. Να το προσδιορίσουμε αυτό. Πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται με, την, ε, με αυτά τα θέματα στην στρατηγική 2020 ε, και με τις επερχόμενες κατευθυντήριες γραμμές. Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια α, ε, επικουρικότητα. Πρέπει να προσδιορίσουμε αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο καλύτερα από ό,τι το κάναμε μέχρι στιγμή. Έπειτα, συντονισμό. Κοινά σημεία αναφορά, benchmarking και ε, συνδυασμό αυτών με τον προπολογισμό. Συνοχή των πολιτικών, ίση μεταχείριση και τα προγράμματα που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα για την δημιουργία θέσεων απασχόληση. Αυτά μπορούμε να τα ψάξουμε περισσότερο και να τα αξιοποιήσουμε ως Ευρωπαίοι εταίροι. Θα συμπεριλάβουμε λοιπόν όλα τα σχόλια από διάφορους ομιλητές, τους νέους, τους χιονικούς εταίρους, τους εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, για να είμαι δίκαιη, θα πρέπει να ξαναδώσω το λόγο, αν επιθυμούν, σε προσώπους των οργανώσεων. Υπάρχει κάποιος που να επιθυμεί να πάρει εκ νέου το λόγο. Όχι, καλυφθήκατε. Έχουν υποθεί όλα. Ο κύριο Καρπιέλο. Δύο λεπτά. Να... απαντήσω στο τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα, ιδίως στην Ευρώπη, όπου υπάρχει όλο μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των αγορών εργασίας στα διάφορα κατημέλη και όπου η κινητικότητα γίνεται ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, είναι σημαντικό, είναι θεμελιώδες να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά όπως είναι οι μαθητείες, οι θέσεις άσκησης και έχουμε νομίζω πολύ καλά εργαλεία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έχουμε και στη στρατηγική του 2020 πολύ θετικά στοιχεία τουλάχιστον στην ε, μορφή που έχουμε δει μέχρι στιγμής για τις θέσεις άσκησης και μαθητείας. Και νομίζω ότι υπάρχει τώρα αρκετή ορμή για να προχωρήσουμε σε κάποιες λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ορμή για να βελτιώσουμε και το επίπεδο των νέων οι οποίοι περνάνε σε μαθητείες και θέσεις άσκησης. Γιατί παρά το γεγονός ότι ποικίλει η κατάσταση από μία χώρα στην άλλη, μία κακή θέση άσκηση όπου κάνει κανείς απλώς φωτοτυπίες για τρεις μήνες, αυτό και τίποτα δεν μαθαίνει, αυτό ισχύει για όλες τις χώρες. Σε αυτό το επίπεδο πράγματι πρέπει να κάνουμε κάτι αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους. Ευχαριστώ. Κύριε Σενικιάλ. Για την διάδραση μεταξύ ευρωπαϊκού επίπεδου και εκπαίδευση των νέων. Εδώ χρειάζεται μεγάλη σύνδεση, διότι όταν κανείς παίρνει έναν μαθητευόμενο μπορεί να περιοριστεί στο να του μαθαίνει να βγάζει φωτοτυπίες και να τον πληρώνει 400 ευρώ, μάλλον έναν ασκούμενο. Ενώ ένα μαθητευόμενο, εδώ είναι τα πράγματα πιο σοβαρά γιατί πρόκειται για πραγματική δοκιμή εργασίας και οι επιχειρήσεις έτσι καταλαβαίνουν καλύτερα πόση σημασία έχει η κατάρτιση των νέων. Πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση, η πρακτική μαθητεία είναι κάτι πολύ θετικό. Στη Γαλλία έχουμε ένα καλό πρότυπο στις ασφαλίσεις. Υπάρχει το παρατηρητήριο των επαγγελμάτων που δηλώνει στις σχολές ποιες είναι οι ανάγκες που υπάρχουν. Τόσοι εμπορικοί εκπρόσωποι, τόσοι κομποτριπούδες, τόσες κομποτριπούδες κλπ. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένοι τομείς όπου δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι νέοι βγαίνουν με το δίπλωμά τους και έχουν 100% απασχόληση από τον πρώτο μήνα. Γιατί υπάρχει αυτή η διάδραση, αυτός ο διάλογος. Πρέπει λοιπόν να συνδέεται το ένα με το άλλο. Η μαθητεία είναι κάτι που μπορεί να διευκολύνει τα πράγματα και επιτρέπει στα σχολεία να, η διασύνδεση να καταλάβουν ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Άρα η σχέση αυτή μεταξύ κατάρτισης και επιχειρήσεων είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πρέπει να ζητήσουμε από τους διάφορους τομείς να οργανώσουν και αυτοί ένα τέτοιο είδους παρατηρητήριο όπου να δηλώνουν τις ανάγκες τους προς τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Να πάρουμε δηλαδή ως πρότυπο αυτό το γαλλικό παράδειγμα γιατί θα μπορούσε να αποτελέσει καλό ευρωπαϊκό πρότυπο έτσι ώστε να βγαίνουν από τα σχολεία νέοι που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης και δεν τραυματίζονται από τις πρώτες τους εμπειρίες. Πάρα πολύ πλούσια ήταν αυτή η ανταλλαγή απόψεων, η οποία μας επιτρέπει να περάσουμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Τούρνεν στη συνέχεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους αυτούς που έλαβαν μέρος στη συζήτηση αυτή και προφανώς Μπορείτε με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνία να επανέλθετε στη συζήτηση με τα μέσα αυτά τα οποία τα γνωρίζετε και τα χρησιμοποιείτε πολύ καλά. 31 Μαρτίου συμφώνησα με την συγγήτρια στι 12 το μεσημέρι να είναι μια κατάθεση τροπολογιών. Και στι 27-28 Απριλίου θα επανέλθουμε στη συζήτηση του θέματο αυτού. Κλείσαμε αυτό το σημείο στη μέση διάταξη και τώρα περνάμε στο 18 που μας οδηγεί στο να αντιμετωπίσουμε για πρώτη φορά την έκθεση πρωτοβουλίας της κυρίας Φιγκυρέντου για το ρόλο του ελάχιστου εισοδήματος στον αγώνα κατά της ένδυας και την προώθηση μια Ευρώπης που βασίζεται στην κοινωνική ενσωμάτωση. Έχουμε ορισμένου προσκεκλημένους. Και σε αυτή την περίπτωση θα σας πρότεινα να δώσουμε το λόγο πρώτα απ' όλα στην εισηγήτρια για να μας κάνει εν συντομία μία εισαγωγή στην έκθεσή της και στη συνέχεια να δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ούτως ή άλλως θα συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει προηγουμένως γιατί οι νέοι εξακολουθούν να είναι και σήμερα θύματα ένδυας για όλους τους λόγους τους οποίους προαναφέραμε. Η ίδια η έννοια της ένδυας όπως ξέρουμε δεν είναι εύκολο να οριοθετηθεί. Εγώ πιστεύω πρέπει να είναι μια πολυδιάστατη αντιμετώπιση στην Ένδια, όχι λαμβάνοντας υπόψη μονάχα τα εισοδήματα, αλλά την κοινωνική ευμάρεια, την πρόσβαση σε απαραίτητες υπηρεσίες, παιδείας, ε, στέγασης, περίθαλψης, δικαιοσύνης, τα θέματα της κοινωνικής προστασίας και ασφάλειας. Πρέπει να έχει αυτή τη μορφή λοιπόν η αντιμετώπιση των νέων ώστε και τα δικαιώματά τους να μπορούν να εφαρμόζονται στην πράξη. Η ένδια είναι ουσιαστικά μία παραβίαση, ένας ακροτηριασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο αγώνας κατά της ένδυας θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν στρατηγικές, ότι υπάρχουν εκπονήσεις σχεδίων μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020. Και όλα αυτά περιλαμβάνουν τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και τις μακροοικονομικές πολιτικές. Λοιπόν, θα ήταν καινοτομία αυτές οι πολιτικές να δίνουν προτεραιότητα στους ανθρώπους και τα, την έξοδο από την ένδια και όχι μονάχα τη σταθερότητα των τιμών. Αυτό θα εξασφάλιζε ότι υπάρχει πραγματική εγγύηση των δικαιωμάτων αυτών των ατόμων, ότι μπορούν να έχουν απασχόληση με ποιότητα, ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις κέρυες δημόσιες υπηρεσίες, ότι έχουν τις απαραίτητες κοινωνικές παροχές, όπως δεν γίνεται σήμερα. Θα σήμαινε ουσιαστικά ότι θα είχαμε μια Ευρώπη πιο δίκαια. Σήμερα που είναι τόσο μεγάλη ανεργία και η επισφαλής και κακοπληρωμένη εργασία αυξάνεται, η ένδια ακόμα και με την στενή έννοια η οποία είναι συζητήσιμη βάσει των τελευταίων στοιχείων θίγει αυτή τη στιγμή πάνω από 85 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι γροθιά στο στομάχι. Μας υποχρεώνει, θα πρέπει να μας υποχρεώσει να κάνουμε στροφή στην πολιτική μας, να έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θέλουμε εμείς να προχωρήσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία για μια έκθεση για την ένδια. Δεν είναι μια έκθεση για ελάχιστα εισοδήματα μονάχα, αλλά μια έκθεση για πολλά είδη ελαχίστων παροχών. Όχι μονάχα στην αμοιβή, στην εργασία, στον εθνικό ελάχιστο μισθό παραδείγματος χάρη. Είναι απαραίτητο να υπάρχει και για τους εργαζόμενους και για τους ασκούμενους είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα ελάχιστο για τις συντάξεις, για τις λεγόμενες κοινωνικές συντάξεις και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν το οποίο χρειάζεται είναι να μιλήσουμε για ελάχιστες παροχές ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι στην κοινωνία μας έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Δεν χρειάζεται να είναι αυτά τα ελάχιστα τα ίδια σε όλες τις χώρες θα πρέπει προφανώς να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο και τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. 500 ευρώ παραδείγματος χάρη ή 475 στη χώρα μου. Σε άλλες χώρες μπορεί να είναι λιγότερο αυτό το ελάχιστο ποσό. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να ε, <clears throat> βασιστούμε μονάχα στο ποσό αυτό. Θα πρέπει να ξέρουμε η υγειονομική περίθαλψη είναι δωρεάν ή πρέπει να πληρώσει κανείς. Θα πρέπει να πληρώνει κανείς για την νοσοκομιακή περίθαλψη. Το ίδιο πράγμα για την παιδεία, το ίδιο πράγμα για τις άλλες ουσιαστικές υπηρεσίε που δίνει το κράτος στον πολίτη. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δούμε το θέμα αυτό υπό το πρίσμα των πολλαπλών διαστάσεων που έχουν οι ελάχιστες παροχές και όχι μονάχα με την στενή έννοια της αμοιβή του επίπεδου εισοδήματος. Αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια νέα πολιτική κατανομής των παροχών και σε μια νέα αντιμετώπιση των ουσιαστικών ε, υπηρεσιών και επίσης και μια νέα αντιμετώπιση για τα πιο εύθραστα κοινωνικά στρώματα όπως είναι οι νέοι, όπως είναι οι γυναίκες γιατί δείχνουν οι στατιστικές ότι το πρόσωπο της ένδυας είναι γυναικείο. Οι περισσότεροι ενδεείς είναι γυναίκες. Είναι γυναίκες είτε νέες είτε ηλικιωμένες που δεν έχουν πρόσβαση σε μια ελάχιστη ανεκτή σύνταξη και που ζουν σε μια κατάσταση ακραίας ένδειας. Επομένως, είναι απαραίτητο να υπάρξουν μέτρα, πολλαπλά μέτρα, ποικίλα μέτρα, για να υπάρξει μια δίκαια ανακατανομή των εισοδημάτων, για να μπορεί να υπάρχει η πρόσβαση όλων αυτών των πιο ευαίσθητων και τροτών στρωμάτων του πληθυσμού, και εδώ μιλάμε για τα άτομα που έχουν αναπηρίες που είναι μετανάστες, τις ατυπικές μορφές οικογένειας. Πρέπει όλα αυτά τα στρώματα του πληθυσμού να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη προσοχή. Και επειδή βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Έτος Αγώνα κατά της Ένδυας, με την έκθεση αυτή θέλουμε να τονίσουμε το ενδιαφέρον και τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προέρθει μια απάντηση στα προβλήματα αυτά που δεν θα είναι απλώς φραστική αλλά θα προσπαθήσει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, θα προχωρήσει στην χάραξη πολιτικών οι οποίες είναι απαραίτητε για να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα των ανθρώπων αυτών που θέλουν να έχουν κάποιο όφελος από όλα αυτά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο στο σύνολό του αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να κάνουμε κάποια μικρή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των ατόμων αυτών και όχι να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση άκρα αδικίας που πλήττει τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Ένδια. Σας ευχαριστούμε για την ε, πρώτη αυτή παρέμβασή σας. Τώρα θα δώσω το λόγο στους τέσσερις προσκεκλημένους μας και στη συνέχεια θα υπάρξει κοινή συζήτηση. Από τους κοινωνικούς εταίρους έχει το λόγο, αλφαβητικά προχωρώ, δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, τον κύριο Άρη Λουρντέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που ε, προσκαλέσατε τις ΣΕΡΕΣ στη συζήτηση. Με άγγιξε πραγματικά αυτό που είπε η προηγούμενη ομιλήτρια, δηλαδή η θέληση του Κοινοβουλίου να δεσμευτεί συγκεκριμένα με μέτρα πιο στεναρά και όχι μόνο με δηλώσει. Γιατί όντως έχουμε πήξει από δηλώσει. Δεν μιλάω για τις δηλώσεις του α, Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στο, α, στον ΟΗΕ, αλλά αν πάρω τη σύσταση του 1992. Ε, βλέπετε, το, το δείχνει και το κεφάλι με τα άσπρα μαλλιά. Ήδη το 1992 συμμετείχε σε αυτή τη συζήτηση τότε. Τι λέγαμε λοιπόν. Αναγνωρίζουμε το θεμελιώδης δικαίωμα ε, στα άτομα για επαρκείς πόρους για να εξασφαλίσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ε, Μιλάω για άτομα τα οποία δεν έχουν θα πέσει του νοικοκυριού τους επαρκείς πόρους κτλ. Ε, αυτές ήταν οι δηλώσεις για το 92. Αρκούν οι δηλώσει. αρκούν οι συστάσεις. Τώρα πρέπει να περάσουμε στις πράξεις, να βρούμε μέσα και εργαλεία για να απαντήσουμε στο πρόβλημα. Είπατε ότι οι αιτίε είναι πολλαπλέ. Διαπιστώνουμε εδώ και πολλά χρόνια ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήσαμε βέβαια θέσεις απασχόλησης, αλλά αυτές οι θέσεις απασχόλησης χαρακτηρίζονται κυρίως από μια βεβαιότητα. Είναι επισφαλής. Ε, ορίστου χρόνου, έκτακτη εργασία, μερική εργασία που δεν την επιλέγει κανείς, που δεν την επιθυμεί κανείς. Φυσικά, αν, δούμε το, αν θεωρήσουμε το ποτήρι είναι μισοάδιο, μπορούμε να πούμε ότι η φτώχεια πριν την κρίση δεν αυξήθηκε ουσιαστικά, αλλά δεν μειώθηκε κιόλας. Μια άλλη επίσημη δέσμευση το 2000 ποια ήταν. Είχαμε δεσμευτεί να εξαλείψουμε υποτίθεται τη φτώχεια. Δεσμευτήκαμε. Η διαπίστωση ποια είναι. Υπάρχει ακόμα φτώχεια. Επιπλέον, οι επισφαλείς εργασίες οι επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Δημιούργησαν φτωχούς εργαζόμενους. 20 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άντρε και γυναίκε, που έχουν θέση απασχόληση. Δεν μιλάμε τώρα για το στάζ, δεν μιλάμε τώρα για τη μαθητεία. Έχουν δουλειά και όμω δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώ από τη δουλειά του. Για τα κεφάλαια τη απασχόληση, οι κοινωνικοί εταίροι έχουν κάνει κάποια πρόοδο στις 9 ε, Δεκεμβρίου του 2009 υπέγραψαν μια συμφωνία, όπως θα ξέρετε, για μια αγορά εργασίας που συμπεριλαμβάνει και, όχι, και δεν αποκλείει τον κόσμο, που τον εντάσσει και δεν τον αποκλείει. Είναι η πρώτη φορά που οι κοινωνικοί εταίροι λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο αυτούς που έχουν δουλειά, αλλά και αυτούς που δεν έχουν, για να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν θέση απασχόλησης. Επί πολύ καιρό είπαμε ότι η απασχόληση είναι ο εγγυητής κατά της του αποκλεισμού και της φτώχειας. Αλλά βλέπουμε ότι πια η απασχόληση δεν είναι αυτή η εγγύηση. Γιατί η σημερινοί φτωχοί εργαζόμενοι θα γίνουν αύριο φτωχοί συνταξιούχοι. Υπάρχει έτσι μία αλυσιδωτή σχέση. Τώρα για αυτούς που δεν έχουν δουλειά. Για διάφορους λόγους. Εμείς τι ζητάμε. Να υπάρξει ήδη από σήμερα ένα μέσο, ένα εργαλείο. Να το συζητήσουμε βεβαίως, αλλά θα εξασφαλίζει θα εξασφαλίζει όχι ακριβώς το ελάχιστο εισόδημα, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Γιατί από την άλλη θέλουμε να ζει ο κόσμος αυτός αξιοπρεπώς και να είναι πολίτης 100%. Γι' αυτό θα εξασφαλίζει ας πούμε ένα εισόδημα. Σήμερα όμως τι γίνεται στα κράτη-μέλη, σε πολλά από τα κράτη-μέλη υπάρχει είτε ένα εισόδημα είτε ένα επίδομα. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν αυτά τα εισοδήματα είναι πάντα κατώτερα από το κατόφλι φτώχειας, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή 60% του μέσου εισοδήματος. Τι σημαίνει έχουμε πρόσβαση σε ένα εισόδημα, όταν αυτό το εισόδημα δεν μας επιτρέπει ούτε καν να φτάσουμε στο κατόφυλλο τη φτώχεια. όχι να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Επομένως, η ΣΕΙΕΣ θέλει όχι μόνο το δικαίωμα στο εισόδημα, όχι το επίδομα, έτσι, το δικαίωμα στο εισόδημα, αλλά το εισόδημα αυτό να υπάρχει για να ζούμε αξιοπρεπώς με βάση όλες τις δηλώσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Αυτό το εισόδημα θα συνοδεύεται από ένα εργαλείο αποτρεπτικό για αυτούς που δεν θέλουν να το εφαρμόσουν. Την περασμένη εβδομάδα είχα πάει σε μια χώρα, δεν θέλω να το κατονομάσω για να μην ε, θυμώσουν διάφοροι. Ε, με είχαν ε, προσκαλέσει συνδικαλιστές α, της χώρας αυτής και υπήρχε και ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης της χώρας αυτής που έλεγε ότι εμείς μιλάμε όχι για εξάλληψη τη φτώχεια, αλλά για μείωση κατά 25%. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη μείωση. Τι θα πει αυτό. Δεν αρκεί η καλή θέληση. Πρέπει να προβούμε σε πράξεις. Ναι, ναι, ναι υπερεύει λίγο το χρόνο μου. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικά και νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεργαστούμε κι εμείς για να υπάρξουν αυτά τα εργαλεία για τα ελάχιστα εισοδήματα. Ευχαριστούμε κύριε Λουρδέλ για την Business for Europe, κυρία Ρεμπέκα Σπίς. Ευχαριστώ Πρόεδρε εξ ονόματος της Business Europe για την πρόσκλησή σας. Εδώ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η δυνατότητα των νέων για να προστατευτούν από τους κινδύνους της οικονομικής ζωής δεν είναι σε καλή κατάσταση εκτός αν εντατικοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις στις διάφορες χώρες μέλη. Η Business Europe για την καταπολέμηση της ανέχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού θεωρεί ουσιώδες στα ευρωπαϊκά κοινωνικά συστήματα να βασιστούν στην αύξηση της απασχόλησης αλλά και της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Η Business Europe έκανε αυτό την τελευταία της δημοσίευση Growth for Europe όπου λέγει να διπλασιαστεί η δυνατότητα ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η οικονομία αν αναπτυσσόταν κατά 2% αντί για 1% δημιουργούνταν εκατομμύρια θέσεων εργασίας. Και για να βγούμε από την κρίση, για να αντιμετωπίσουμε τις δημογραφικές αλλαγές και να καταπολεμήσουμε την ανέχεια και την κοινωνικό αποκλεισμό πρέπει να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της σταθεροποίησης των ε, δημοσιονομικών αγορών, των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ορισμένα σχόλια τώρα για, το, για τη στρατηγική της Ένωσης για το 2020 και μετά. Εμείς θεωρούμε ότι η στρατηγική αυτή είναι χρήσιμη βάση για την ανάπτυξη μιας πιο δυνατής Ευρώπης, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν όλα αυτά πιο γρήγορα. Και όπως υπόθηκε σωστά, πρέπει για να καταπολεμηθεί η ενεργεία των νέων να καταπολεμηθεί και η ανέχεια και να βελτιωθούν τα συστήματα κοινωνικής περίθαλψης. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η ασφαλιξία είναι τμήμα της στρατηγικής αυτής. Μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων επίσης για να μπορούν να εργάζονται με τρόπο πιο ευέλικτο στην αγορά εργασίας. Βέβαια η Business Europe υποστηρίζει την διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμησης της, της Ανέχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού που θα τελειώσει μένει το 2010 αλλά θα έπρεπε να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και θεωρούμε ότι η βιωσιμότης και η κοινωνική περίθαλψη καθώς και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε όλες τις υπηρεσίες είναι ουσιώδης παράγοντες για την καταπολέμηση της ανέχειας και του ελληνικού αποκλεισμού. Για την αγορά εργασίας συγκεκριμένα η Business Group θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η απασχόληση είναι βασικό δικαίωμα και προτεραιότητα πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο απασχολησιμότητας αν θέλουμε να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη και διατήρηση των συστημάτων κοινωνικής περίθαλψης. Όπως ξέρουμε και από την κρίση, όπως μάθαμε από την κρίση, έχουν υπάρξει ορισμένες επιτυχείς μεταρρυθμίσεις για πιο ευέλικτη τη οργάνωση του χρόνου εργασίας α πούμε και αυτό δημιουργεί και αυτό θέσει εργασίας. Δημιουργεί το σωστό πλαίσιο για την ε, μείωση του κόστου της εργασίας. Κατά τις προβλέψεις του ΣΑ μπορεί να αυξηθεί η απασχολήση κατά 0,6% ήδη από φέτος. Βέβαια τα συστήματα περίθαλψης πρέπει να στηρίζουν τα εισοδήματα και των ανέργων, αλλά κυρίως να τους σωθούν να βρουν μια νέα θέση εργασίας. Αυτό το έχω πει και άλλες φορές και για την ασφαλιξία και τις αρχές της, τη διαβίωμα μάθηση και τα λοιπά, όλα τα έχω πει. Όπως είπε και η συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, εμείς στους κοινωνικούς εταίρους έχουμε αναλάβει δράσεις στον τομέα αυτών, δημιουργώντας μία συμφωνία πλαίσιο για τη σφαιρική αγορά εργασίας. Και αναγνωρίζουμε ότι πρέπει για να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή και ανάπτυξη από κοινού οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες να αναλάβουν πρωτοβουλία. Η συμφωνία αυτή στοχεύει ιδιαίτερα σε εκείνου που έχουν δυσκολίες όχι μόνο εισόδου στην αγορά εργασίας αλλά και στη συμπερίληψή τους σε αυτήν. Για το ελάχιστο εισόδημα φυσικά συμφωνούμε ότι είναι προτεραιότητα και αυτό για την αξιοπρέπεια του εργαζομένου. Πρέπει όμως να εξισορροπηθούν οι ανάγκες του κάθε ατόμου με το κοινωνικό σύστημα ώστε να μπορεί ο καθένας να ζει αξιοπερεπώς. Σχεδόν όλες οι χώρες μέλη έχουν προβλέψει κάτι εθνικά για το στόχο αυτόν, αλλά αυτό είναι βραχυπρόθεσμο. Η έκθεση τονίζει επίσης τις διαφορές που έχουν τα εθνικά προγράμματα και Σωστά λέγεται ότι ο στόχος πρέπει να είναι να μην υπάρχουν αντικίνητρα για την εξέβρεση εργασίας από τις προτάσεις αυτές. Τέλος, για την εφαρμογή των προτάσεων αυτών, πιστεύουμε ότι ο συντονισμός και η συνεργασία είναι παραμένουν ο καλύτερη μέθοδος για την επιτυχία και καλύτερη μέθοδος είναι μια περιοδική αναθεώρηση των όλων των ενδιαφερομένων. Ευχαριστώ πολύ. Τελεία. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσουν τώρα οι εκπρόσωποι. Ο κύριος Φίντον Φάρελ πρώτα από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης της Ανέχειας. Έχετε το λόγο κύριε Φάρελ μου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι αργά. Αλλά παρόλα αυτά να σας ευχηθώ καλή μέρα του Αγίου Πατρικίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που στέφει την προσοχή του σε αυτό το θέμα και αναγνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια το Κοινοβούλιο έχει εκπονήσει σημαντικές εκθέσεις για αυτό το σημείο. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε την προσπάθεια. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος του ΣΕΡΕΣ της ETUC, θα πρέπει να γίνουν και βήματα προς τα εμπρός. Όχι να επαναλάβουμε αυτά που κάναμε στο παρελθόν. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω από των προτέρων ότι είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε για να προχωρήσετε. Ε, υπάρχει η σύσταση αυτή για την ε, ενεργό ένταξη. Ε, τώρα είμαστε στο επόμενο βήμα. Ε, υπάρχει η έκθεση Fraser και Marlier για τα, ελάχιστα, για τα προγράμματα ελάχιστων εισοδημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθούμε να αναπτύξουμε και δείκτες για την ενεργό αυτή ένταξη. Ελπίζω αυτή η έκθεση να υποστηρίξει την προηγούμενη δουλειά που σας ανέφερα, οι δουλειές. Ελπίζω όλες οι πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο να εξασφαλίσουν ότι αυτή η έκθεση θα δυνατή, στεναρή και ζητώ από την εισηγήτρια να το εξασφαλίσει αυτό. Το δικαίωμα σε ένα ελάχιστο εισόδημα είναι ένα θεμελιώδες εισόδημα και είναι σημαντικό για να μπορέσει να ζήσει κανείς αξιοπρεπώς, να υπάρχει ένα τέτοιο εισόδημα. Δεν ξέρω πόσοι από εσά το χρησιμοποίησατε. Εγώ στη δική μου ζωή το χρειάστηκα και πραγματικά σημείωσε διαφορά. Μπορεί να μην ήταν επαρκές, αλλά το γεγονός ότι μου δόθηκε κάτι ήταν σημαντικό για να με κρατήσει σε σχέση και σε φάση με την κοινωνία. Θέλω να τονίσω λοιπόν τη σημασία αυτών των προγραμμάτων, γιατί πραγματικά υπερασπίζουν θεμελιώδη δικαιώματα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην γενικεύουμε πολύ και να αναγνωρίζουμε το ρόλο αυτού που συζητάμε. Το κλασικό πρόγραμμα ε, ελάχιστου εισοδήματο είναι ένα πρόγραμμα που αφορά ανθρώπου που είναι διαθέσιμοι για να δουλέψουν, αλλά δεν βρίσκουν δουλειά. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλους όσους βρίσκονται σε παρόμοιε συνθήκες. Ε, ακούσαμε για το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου αυτό το ελάχιστο εισόδημα δεν υπάρχει σε, για ανθρώπους που είναι κάτω των 25. Αυτό είναι απαράδεκτο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε την ιδέα της επάρκειας του ελάχιστου εισοδήματος για να καλύπτει και την, τις μετέπειτα φάσεις της ζωής μας. Παραδείγματος χάρη και την επάρκεια των συντάξεων και των οικογενειακών επιδομάτων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια σφαιρική εικόνα η έκθεση μιλάει για το ρόλο του ελάχιστου εισοδήματο για την καταπολέμηση τη φτώχεια και τη ένταξη στην κοινωνία. Έτσι, καταρχάς, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι το βασικό εργαλείο για την πρόληψη και την ελάφρυνση των επιπτώσεων της φτώχειας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν τη σημασία του προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Εγώ συνεργάστηκα πολύ με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήταν πολύ μακριά από την εργασία και ήταν αποκλεισμένοι. Ε, δεν είναι δύσκολο να τους κινητοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους για να προχωρήσουν προς την αγορά εργασίας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν τα μέσα. Και αυτό το ελάχιστο εισόδημα είναι ένα μέσο για να τους κρατήσει σε επαφή και να τους δώσει τα κίνητρα για να κάνουν ένα βήμα προκειμένου να βρουν τελικά μια αξιοπρεπή εργασία. Το... Επίσης, αυτά τα προγράμματα είναι οικονομικοί ε, σταθεροποιητές, όχι μόνο για τα άτομα που είναι αποδέκτες αλλά προστατεύουν και την ίδια την κοινωνία και την καθιστούν δυνατή. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης και με αυτή την έννοια το ρόλο που παίζει το πρόγραμμα ελάχιστου εισοδήματος. Επίσης... Ξέρουμε επίσης ότι τα συστήματα αυτά για ελάχιστο εισόδημα μπορούν να είναι χρήσιμα στο να αναπτύξουν μεγαλύτερη ισότητα σε μια κοινωνία. Ξέρουμε ότι οι κοινωνίες με ισότητα λειτουργούν καλύτερα για όλους ακόμα και για τους φτωχούς. Νομίζω ότι αρχίζουμε επομένως να περνάμε το μήνυμα για τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ευνοεί το σύνολο της κοινωνίας και μονάχα όχι τους φτωχούς. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα αρνητικά στερεότυπα που έχουν να κάνουν με το θέμα αυτό των συστημάτων ελαχίστου εισοδήματος που νομίζουν πολύ ότι αυτό αφορά μονάχα τους φτωχούς. Έχω κάποιες πολύ λεπτομεριακές προτάσεις αλλά το έγγραφό μου θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέλη της Επιτροπής γιατί δεν έχω το χρόνο να τα συζητήσω όλα αυτά τα θέματα. Είναι σημαντικό πάντως να πούμε ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα για να δούμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελαχίστων εισοδημάτων. Ξέρουμε ότι το 60% του μέσου εισοδήματος είναι ένα πολύ καλός, ένας πολύ καλός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το τι είναι επαρκές αν το εισόδημα ή όχι και έχουμε χρησιμοποιήσει τις στάνταρτ μεθοδολογίες για να δούμε τι ακριβώς χρειάζεται, γιατί όπως είπε και η η Ρέντο, η αποτελεσματικότητα συνδέεται όχι μονάχα με το χρηματικό εισόδημα, αλλά και με την πρόσβαση σε άλλες μορφές υπηρεσίες και με την υποστήριξη για να μπορεί να υπάρχει μια απασχόληση ποιότητας. Αυτό το οποίο είναι ουσιαστικό για μας που ζητάμε σε αυτή την έκθεση είναι να ζητήσετε να υπάρχει μια οδηγία πλαίσιο σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελαχίστου εισοδήματο και έχουμε συγκεκριμένε προτάσει για το τι θα μπορούσε να είναι το περιεχόμενο μια τέτοια οδηγία. Δεν είναι μια πανάκια που θα καλύψει όλα τα θέματα με ένα ενιαίο τρόπο, αλλά ένα πλαίσιο για να μπορέσει το κάθε κράτος μέλος να αναπτύξει τα δικά του συστήματα. Είναι μια διαδικασία που μπορούμε να σας δώσουμε τις κατευθυντήρες γραμμές και το σκελετό για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να το αναγνωρίσετε αυτό στην έκθεσή σας. Έχω καταδαπανίσει πολύ χρόνο. Θέλω απλώς να επαναλάβω <clears throat> ότι αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι να υπάρχει μια πραγματική συνέχεια στην σύσταση για ε, ελάχιστες αποδοχές να υπάρχει πραγματική παρακολούθηση αυτής της σύστασης για ελάχιστες αποδοχές και να εξασφαλίσουμε φυσικά ότι αυτή η έκθεσή σας με τον τρόπο αυτό, με τη σύσταση για μια οδηγία πλαίσιο για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελαχίστων εισοδημάτων είναι, είναι θετική. Κλείσαμε με αυτά που είχαν να μας πούν οι καλεσμένοι μας και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην συζήτηση. Α συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, συγχωρείτε. Η κυρία Ντιπούπο έχει το λόγο. Από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πλατφόρμα. Με συγχωρείτε, συγγνώμη, έχετε έξι λεπτά κι εσείς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω ζητήσει από τα παιδιά μου να έρθουν εδώ σήμερα από την Τετάρτη απόγευμα και αυτό ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας και τα ευρωπαϊκά δίκτυα για τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε ένδια, τους φτωχού, τις γυναίκες, τους νέους. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια συνένεση για το πόσο σημαντικό είναι το ελάχιστο εισόδημα και πόσο σημαντικό είναι αυτό το εργαλείο. Εμείς θέλουμε πραγματικά να γίνει κάτι τέτοιο και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι υπάρχει τώρα μια έκθεση που την προετοιμάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Πέντε μηνύματα θέλω να σας δώσω. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να επανέλθουμε στον αρχικό στόχο. Ποιο είναι το επίπεδο δεσμευσή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αναχαιτήσουμε την ένδια και τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα γιατί η, το ελάχιστο εισόδημα είναι ένα εργαλείο αλλά το ερώτημα είναι κατά πόσο εξυπηρετεί πλήρως το στόχο μας, ο οποίος στόχος είναι να αντιμετωπίσουμε την ένδυα στην Ευρώπη. Έχουμε 80 εκατομμύρια φτωχούς στην Ευρώπη. Είναι μια ολόκληρη Γερμανία. Ένα παιδί σε κάθε πέντε ζει σε ένδυα. Θέλουμε ακόμα να το εξαλείψουμε αυτό ή όχι. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ θετικό μήνυμα επίση από τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 που λέει ότι ένα από του πέντε κύριου στόχου για την επόμενη δεκαετία θα πρέπει να είναι η εξάλληψη τη ένδυα στην Ευρώπη. Είναι ένα πολύ σημαντικό θετικό βήμα γιατί σε μια κοινωνία δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει αν δεν συνδυάσει το θέμα της καινοτομία, της οικονομικής πρόοδου, αλλά και της εξάλληψης ή τουλάχιστον του περιορισμού της ένδυας. Αυτή τη στιγμή η πρόταση που έχουμε εμείς από την Κομισιόν έχει ένα συγκεκριμένο στόχο και ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα επιμείνει σε αυτό το στόχο της Κομισιόν γιατί το θέμα αυτό θα συζητηθεί και από το Συμβούλιο στο τέλος του μήνα και θα ήθελα και το Κοινοβούλιο να επιμείνει για τους στόχους της ε, μείωσης ένδυα και να υποστηρίξει του δείκτε οι οποίοι συνδυάζονται με αυτή την πολιτική στα πλαίσια τη πρότασης τη Κομισιόν. Το επόμενο σημείο είναι, το επόμενο μήνυμα είναι όταν έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο να ξέρουμε ποια είναι τα εργαλεία τα οποία θα είναι αποτελεσματικά. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι το ελάχιστο εισόδημα. Όπω είπε η κυρία Φιγκερέντο, η πρόσβαση στι δημόσιε υπηρεσίε, η υγειονομική περίθαλψη, επαρκή συντάξει κτλ. <clears throat> Ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Το έχουμε κάνει εδώ και πολύ χρόνο. Ξέρουμε λοιπόν ότι μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο και έχει μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν η ένδυα στην Ευρώπη. Τώρα δυστυχώ λόγω της κρίσης δεν υπήρξε αναγνώριση του ρόλου των κοινωνικών σταθεροποιητών. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας πραγματικά βοηθούν τους ανθρώπους να ξεπεράσουν την κρίση και τα συστήματα ελαχίστου εισοδήματο μπορούν να διατηρήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο κατανάλωση μεταξύ του πληθυσμού. Αυτό είναι το δεύτερο μήνυμά μου προ εσά, μέλη του Κοινοβουλίου. Πώ μπορούμε να μην αναφερόμαστε στα θέματα των κοινωνικών σταθεροποιητών σε ένα καιρό κρίση. Αναφέρθηκε πέρσι το θέμα αυτό και τώρα πάλι το ξεχάσαμε. Και πάλι δεν υπάρχει αρκετή ορατότητα αυτών των δικτών να τονίσουμε πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι δείκτες για την βιωσιμότητα στις κοινωνίες μας. Θα πρέπει να τονίσουμε λοιπόν το ρόλο των συστημάτων κοινωνικής προστασίας σαν ένα βασικό κεφάλαιο της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αυτό είναι το δεύτερο μήνυμα που έχω να κάνω σε σχέση με την έκθεση και το ρόλο σας. Το τρίτο σημείο που θέλω να θίξω αφορά τις συνθήκες εργασίας και το αναφέραμε προηγουμένως. Νομίζω ότι κάτι το οποίο μας ανησυχεί πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι όταν επιδεινώνται οι συνθήκες εργασίας έχει και άλλο αντίκτυπο σε αυτούς που ζουν με ένα ελάχιστο εισόδημα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και πιο επισφαλείς θέσεις Τα άτομα αυτά δεν έχουν ε, επιδόματα ανεργίας όταν χάνουν τη δουλειά τους και καλύπτονται μόνο από τα συστήματα αυτά ελαχίστου εισοδήματος όταν υπάρχουν όλα αυτά τα νέα συστήματα που λένε ότι ο άνεργος θα πρέπει να ψάχνει να βρει μια θέση εργασίας. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τελικά μειώνεται το εισόδημα των ατόμων, οι οποίοι αναγκάζονται να ψάχνουν όλο και πιο κακοπληρωμένες δουλειές. Και επομένως δεν λειτουργεί το σύστημα, δεν βγαίνει κανείς με την εργασία από τον χώρο της ένδυας. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρξει μια ελάχιστη ποιότητα της ε, απασχόλησης για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα αυτό του ελαχιστού και υπάρχει επίση και ο αρνητικό τρόπο παρουσίαση για αυτού οι οποίοι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά επιδόματα. Του θεωρούν ότι είναι εγκληματίες ή απαταιώνε, ότι πρέπει να βρει κάποιο μια δουλειά για να έχει εισόδημα. Τα άτομα αυτά λοιπόν τα οποία δεν έχουν τα λεφτά να ζήσουν θεωρούνται ότι κάνουν κατάχρηση του συστήματο. Εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί όλα συνδέονται. Και το τρίτο μήνυμα είναι ότι καλωσορίζουμε την έκθεση αυτή για την ποιότητα της απασχόλησης. Λυπόμαστε γιατί η στρατηγική Ευρώπη 2020 δεν ήταν ένας από τους βασικούς στόχους. Νόμιζα ότι υπήρχε συνένεση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά όχι ποιοτικών θέσεων. Και δεν υπάρχει καν αυτό το θέμα ε, και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020. Το τελευταίο θέμα είναι για την ισότητα. Ε, κυρία Φιγκερέιδο, είπατε κάτι πολύ σωστό θα πρέπει να δούμε διάφορες ομάδες ε, στην κοινωνία που δεν επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο. Οι γυναίκες, Φερρυπίν. Έχουμε πολλέ μητέρες μόνες με παιδιά που ζουν σε συνθήκε φτώχεια. Και εδώ μπαίνει το θέμα της ποιοτική θέση απασχόλησης. Ε, αν θες να επιβιώσεις, δεν αρκεί ένα εισόδημα. Ε, άμα έχεις και παιδιά, δηλαδή, πρέπει να έχεις οπωσδήποτε δύο πηγές εισοδήματος. Και αυτό πρέπει να το, λάβουμε υπόψη μα, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία με διαζύγια κτλ. Ε, υπάρχουν πολλέ δηλώσει. Θα πρέπει να σκεφτούμε τώρα τι οδηγίε. Η οδηγία κατά των, διακρίσεων, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικά. Ο κόσμο ε, εστιάζει την προσοχή του με, σε τέτοια μέσα, όπω οι οδηγίες. Ε, πάμε τώρα στη γενική συζήτηση και θα δώσω το λόγο στην κυρία Λίν. Ε, σας καλωσορίζω όλους. Ε, με ε, γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε συνεργαστεί για αυτό το θέμα. Το 2007 είχα εγώ μία, εκπονήσει μία έκθεση ε, και μιλούσα τότε για το αξιοπρεπές ελάχιστο εισόδημα. Βλέπουμε ότι τα ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια και ότι δεν υλοποιούμε του στόχου μα. Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση, νομίζω, μεταξύ του ελάχιστου εισοδήματο και του ελάχιστου μισθού. Και ξέρω ότι με την πάροδο των ετών ε, ο κόσμο τα έχει μπερδέψει αυτά τα δύο. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για αξιοπρεπές ή επαρκές ελάχιστο εισόδημα, καθώ και ελάχιστο μισθό. Είναι τελείω διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο. μιλήσατε προηγουμένως ο εκπρόσωπος ειδικά ε, του δικτύου για τη φτώχεια ε, για το συντονισμό. Ε, και ο εκπρόσωπος ο άλλος μίλησε για την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Θα ήθελα να μου πείτε, πιστεύετε ότι θα έχει καταφέρει καλά αυτή η μέθοδο συντονισμού για να πετύχει το ελάχιστο εισόδημα. Ε, γιατί δεν ξέρω αν έχει πετύχει τίποτα για τις κοινωνικές υποθέσεις. Πρέπει να αναγνωρίσουμε νομίζω ότι δεν έχει αποδώσει όπως θα περιμέναμε. Ε, και το θέμα είναι πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό το σύστημα να λειτουργήσει καλύτερα. Έπειτα, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να είναι πολύ επιτακτικό. Ε, δεν θα πρέπει να επιβάλλει τα ίδια πράγματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Συμφωνώ. Αλλά ίσως τώρα στο βαθμό που δεν λέμε στα κράτη-μέλη πρέπει να πληρώσετε αυτό το συγκεκριμένο ελάχιστο εισόδημα, στο βαθμό που έχουμε ένα πλαίσιο, νομίζω ότι μπορούμε να κινηθούμε μέσα σε αυτό, Κάλιστα. Τώρα, με αυτό δεδομένο, μιλήσατε για την οδηγία κάτω των διακρίσεων, που έχει κολλήσει στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να μου πείτε όλοι σας, αν βλέπετε να υπάρξει στο μέλλον κάποια οδηγία για το ελάχιστο εισόδημα. Και αν προωθηθεί μια τέτοια οδηγία, τι υποστήριξη θα υπάρχει από το Συμβούλιο, θα κολλήσει και αυτή όπως η οδηγία κατά των διακρίσεων. Και η οποία φαίνεται ότι και για το εγγύς μέλλον και για το προβλεπόμενο μέλλον θα παραμείνει κολλημένη αυτή η οδηγία. Αν ζητήσουμε μια οδηγία πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι παράλληλα με αυτή την οδηγία υπάρχει και κάτι άλλο. Παραδείγματο χάρη η ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Να μην περιμένουμε εξαρτημένοι από το Συμβούλιο να κάνει την αποφασιστική κίνηση ε, αφού εκπονήσουμε τη δική μας νομοδότηση. Αυτά και ευχαριστώ όλους για την ε, ε, συμμετοχή σα και τι παρεμβάσει σα. Ο κύριος Κοφεράτη παρατηρήσεις της κυρίας Φιγκερέιδο είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες. Ε, ας κάνουμε τώρα ένα βήμα προς τα πίσω και να μην ξεχνάμε το θέμα το οποίο συζητάμε είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει εδώ και καιρό και αναφιβόλως επιτάθηκε τα δύο τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Και επειδή στον ορίζοντα δεν διαφαίνονται έτσι γρήγορες ε, βραχυπρόθεσμες ε, λύσεις. Λόγω των δυσκολιών που δημιουργήθηκαν λόγω της κρίσης σε όλα τα κρατημέλη. Γι' αυτό λοιπόν για μεθοδοτικούς λόγους θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα ε, με τρόπο κατεπήγοντα. Και να λάβουμε υπόψη μας ότι ναι μεν κινούμαστε όλοι στο ίδιο πλαίσιο αλλά υπάρχουν και διαφορές. Τώρα, αν δεν υπάρξει γρήγορη ανάπτυξη και αν δεν υπάρξει ανάπτυξη που δημιουργεί νέο πλούτο, τα προβλήματα που αφορούν την κοινωνική προστασία θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα να τα διαχειριστούμε. Τα κράτη θα έχουν λιγότερους πόρους και θα μπουν σε σύγκρουση οι διάφορε ανάγκε των διάφορων ομάδων πληθυσμού. Η απόλυτη προτεραιότητα είναι η στρατηγική 2020 να ξαναβάλει σε κίνηση τις ευρωπαϊκές οικονομίες γρήγορα και να υπάρξουν πιο απτά αποτελέσματα από αυτά που, χάρη, και χάρη σε αυτή τη στρατική από αυτά που θα είχαμε με τρόπο αυθόρμητο. Τώρα, μετά από αυτά, πρέπει να δώσουμε προσοχή και να στραφούμε λίγο στα άτομα τα οποία, για τα οποία μιλάμε εδώ και τα οποία θέλουμε να καλύψουμε με αυτά τα μέσα. Νομίζω ότι καταρχάς αυτό που θα αυξηθεί λόγω της κρίσης είναι η ανεργία και η φτώχεια λόγω της έλλειψης εργασίας. Τα άτομα τα οποία θέλουν να εργαστούν δεν έχουν δουλειά. Και γενικά σήμερα βοηθούνται ενώ βγαίνουν από την επαγγελματική δραστηριότητα και μπαίνουν ως άνεργοι στο ράφι. Και όταν δεν έχουν δραστηριότητα δεν έχουν πολλά εργαλεία στα χέρια τους. Ο ελάχιστος ε, μισθός, όχι το εισόδημα που είναι κάτι άλλο, ο ελάχιστος μισθός μπορεί να γίνει το βασικό εργαλείο για να υπάρξει ομοιομορφία στην υπεράσπιση των πλέον εκτεθειμένων ατόμων. Καταρχά, οι νέοι που δεν είχαν ποτέ δουλειά και θα ήθελαν και τα άτομα τα οποία θέλουν να δουλέψουν και έχουν χάσει τη δουλειά του. Η κατάσταση στα κράτη-μέλη είναι εντελώ ανώμια. Ορισμένοι έχουν κάνει επενδύσεις στους ε, κοινωνικούς ε, σταθεροποιητές, αλλά δεν έχουν επενδύσει όλοι στους ανθρώπινους πόρους όταν αυτοί βρίσκονται σε περίοδο αδράνειας. Νομίζω ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Να υπάρξουν κάποια εργαλεία για όλα τα κράτη-μέλη, διαφθορτικά αποτελεσματικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί το, το, ο αριθμό των ατόμων που, τα ενδιαφέρουν αυτά τα εργαλεία, που ενδιαφέρονται από αυτά τα εργαλεία αυξάνεται από μέρα σε μέρα. Έπειτα, για τα άτομα τη γενιά μου, ο φτωχό ήταν ένα άτομο το οποίο δεν δούλευε. Σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σήμερα αλλάζουν τα πράγματα. Σήμερα υπάρχουν άτομα τα οποία δουλεύουν, κυρίω γυναίκε, και που από τη δουλειά του δεν αντλούν ένα επαρκέ εισόδημα για να ξεπεράσουν το κατόφλι της φτώχειας. Ο όρος φτωχός είναι, ενδεής είναι μια δύσκολη λέξη. Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο εργαζόμενος, ο εργαζόμενος προέρχεται όπου η φτώχεια, ε, από, μια, ε, από ένα περιβάλλον όπου η φτώχεια λόγω του χαμηλού εισοδήματος υπήρχε ήδη. Τώρα, αυτός ο φαύλος κύκλος σπάει μόνο με επενδύσεις στην ε, κατάρτιση. Αλλιώ δεν υπάρχουν αποτελέσματα που μπορούν να απελευθερώσουν αυτά τα άτομα από την ε, δουλειά. Το άλλο, είναι, το άλλο θέμα είναι οι ηλικιωμένοι. Οι ηλικιωμένοι. Οι ηλικιωμένοι είναι φτωχοί γιατί δεν έχουν πια το οικογενειακό εισόδημα, αλλά παραμένουν μόνοι του, ζουν πια μόνοι του. Ε, όταν μιλάμε για το welfare, για το κράτο πρόνοια, θα πρέπει να μιλήσουμε για την ποιότητα ε, του κράτου ε, πρόνοια. Όχι μόνο για τη διάδοσή του, ε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους ηλικιωμένους. Για πολλούς ηλικιωμένους, ίσως η μόνη οδός είναι ε, το κοινωνικό κράτος με παροχές ποιοτικέ και ε, προσαρμοσμένες για να σου εξασφαλίσει ένα επίπεδο ζωής. Ευχαριστώ ο κύριος Χίγγινς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα επειδή μας πιέζει και ο χρόνος δεν ξέρω ποιον ακριβώς εκπροσωπεί η Business Europe, Europe σε ό,τι αφορά επιχειρηματικούς φορείς. Γνωρίζω όμως ποια είναι η πραγματικότητα ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι μεγάλες επιχειρήσεις υποστηρίζουν το να υπάρχει ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Το, το αρνούνται και αρνούνται να υπάρχει ένα ελάχιστο εισόδημα το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων, ιδίως λόγω της ε, παγκόσμιας κρίσης που αντιμετωπίζει ο καπιταλισμός. Το επιχείρημα στην πραγματικότητα είναι ότι θα πρέπει να μειωθούν οι ελάχιστες καταβολές. Αυτό τονίστηκε πάρα πολύ στην Ιρλανδία από τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και λένε επίσης ότι και οι ελάχιστες αμοιβέ, οι ελάχιστοι μισθοί για τους εργαζόμενους θα πρέπει να περικοπούν. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Θέλουν να μειώσουν τις ε, παροχές ε, κοινωνικού χαρακτήρα και συγχρόνω να μειώσουν και τις αμοιβέ. Και αυτό έχει γίνει στην Ιρλανδία. Έχουν μειωθεί και οι μισθοί και οι συντάξει. αλλά συγχρόνω μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα hedge funds, τα διάφορα επενδυτικά ταμεία, κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό οδήγησε σε χάος στην Ελλάδα, όπου η ελληνική κυβέρνηση, κάτω από την πίεση των επενδυτικών ταμείων, αναγκάζεται αυτή τη στιγμή να καταπιέζει τους φτωχούς και τους εργαζόμενους και να περικόπτει τις αποδοχές τους στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα καλά λόγια δεν πρόκειται να αλλάξουν τίποτα. Αυτά λοιπόν κυρία Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σημαντικά για το θέμα των συντάξεων. Σίγουρα, όταν κάποιος έχει περάσει όλη του την ζωή να εργάζεται, η ιδέα μιας αξιοπρεπούς ε, σύνταξης και το να μπορεί κανείς να φεύγει σε μια λογική ηλικία από το χώρο εργασίας, είναι πιστεύω μια βασική ιδέα. Αλλά αυτή η βασική ιδέα πολιτισμού αυτή τη στιγμή υπονομεύεται ε. από τις επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις τι λένε να εργάζεται κανείς ως τα 68 στην Ιρλανδία. Πρέπει δηλαδή οι εργαζόμενοι να πέσουν νεκροί ενώ δουλεύουν για να μην κοστίζουν τίποτα. Μετά αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Και οι συνδικαλιστικοί φορείς, η ETUC και οι άλλοι φορείς κάνουν τις εκκλήσεις τους στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν. Φοβάμαι όμως ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο εμφορούνται πλήρω από την δεξιά νεοφιλελεύθερη ιδεολογία που υποστηρίζει τι επιχείρησει. Μόνο με την κινητοποίηση των εργαζομένων και των φτωχών θα μπορέσει να σταματήσει αυτή η τάση προς όλο και μεγαλύτερη χρήση επισφαλούς εργασίας και μείωση των ε, βιωτικών επιπέδων των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο ενδεχομένως. Και μήπως αν όχι, τότε ένα λεπτό στον καθένα, που δεν θέλει να λάβει το λόγο, των ομιλητών για να καταλήξει επί της έκθεσης Φιγκερέιντο και μετά και η ίδια. Λοιπόν, με την ίδια σειρά, Άρνης Ρόντερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καθησυχάζω τον κύριο Χίγκινς εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα φιλελεύθερος. Εμείς ζητάμε ποιότητα της απασχόλησης. Και κάτι άλλο για το οποίο θέλω να επιμείνω γιατί με ανησύχησε. Έγινε λόγος εδώ η διπλανή μου. Το ήξερα όμως, ξέρω αυτές τις θέσεις. Για μείωση των εισφορών ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Μα η μείωση των εισφορών ποτέ δεν δημιουργήσε απασχόληση. Είναι σαν δώρο στους εργαδότες αλλά δεν δημιουργεί απασχόληση και μειώνει τα έσοδα τα φορολογικά έσοδα και γενικώ τα έσοδα που χρειάζονται ακριβώς για να υπάρξει ένα εισόδημα καλύτερο από το ελάχιστο. Εμείς δεν μιλάμε για ελάχιστο εισόδημα αλλά για αξιοπρεπές εισόδημα. Για να προσέχουμε εδώ. Να μην δίνουμε στον ένα για να τα πάρουμε από τον άλλο. Λοιπόν. Εγώ πάντοτε θυμώνω και ταράζομαι όταν ακούω λόγο, γίνεται λόγος για τέτοια πράγματα όπως μείωση των εισφορών. Πρέπει να βρεθούν νέοι πόροι, νέα μέσα, όπως έγινε για τις τράπεζες. Ε, επ' αυτού είμαι στεναρότατος. Ευχαριστώ κύριε Ρεβέκα Σπίτ. Αφού έχουμε μόνο ένα λεπτό θα απαντήσω στο σχόλιο που μου απευθύνθηκε άμεσα για να αποσαφινιστούν τα πράγματα. Έχουμε 40, εκπροσωπούμε 40 εθνικές ομοσπονδίες και 20 εκατομμύρια μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. μεσαίων και μεγάλων μάλλον. Και από ό,τι έχω δει εγώ, εμείς δεν ζητάμε κατώτατο μισθό, δεν ξέρω από πού το βρήκατε. Εμείς ζητάμε εξισορρόπηση μεταξύ της διατήρησης και συντήρησης των δημοσίων δαπανών οι οποίες έχουν ξεπεραστεί κατά τρομερό επίπεδο και από την άλλη αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής περίθαλψης. Δεν λέμε όχι στο, στο ελάχιστο εισόδημα, αλλά είναι ζωτικό όπως υπόθηκε και από την έκθεση, η έκθεση φέτος, ότι πρέπει να μπορέσουν οι άνεργοι να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας ώστε να υπάρξουν περισσότερα έσοδα για τα συστήματα περίθαλψης. Εκτός αυτού αναφέρατε την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλό εργαλείο για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ χωρών αλλά απ' την άλλη πρέπει να ενισχυθεί η μέθοδος αυτή. Δεν έχω κάνει καμία πανάκια να προτείνω, αλλά θα μπορούσαμε να το ξανασκεφτούμε γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλό εργαλείο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φουνταμπά. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα δεν θεωρούμε ότι απέτυχαν τα συστήματα αυτά. Πετύχανε κάτι και οι προσπάθειε αυτέ κράτησαν ζωντανέ συζητήσει όπω η ενεργή ενσωμάτωση κτλ. Δεν χάσαμε την πολιτική μα ορμή στην αναθεωρημένη ατζέντα τη Λισαβόνα. Ο στόχο τώρα που επιζητείται από τι προτάσει τη Ατζέντα 2020 θα μπορούσαν να δώσουν και πάλι την πολιτική ορμή σε μια στρατηγική αντιμετώπιση τη ένδυα. Αυτό όμως τώρα το οποίο απαιτείται να δημιουργήσουμε κάποια υποστήριξη για την οδηγία πλαίσιο για ένα ελάχιστο εισόδημα και αυτό πρέπει να είναι και ένα αποκοίημα της αντιμετώπισης του έτους 2010 ως έτους κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της ένδυας. Πρέπει να δούμε και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για όλα αυτά. Και τις δύο πλευρές. Τα χρήματα που πληρώνονται για την κοινωνική προστασία ξαναγυρίζουν αμέσως στην οικονομία. Δεν είναι δαπάνη. Είναι επένδυση λοιπόν τα χρήματα αυτά. Δεύτερον, Πρέπει να είναι επαρκή η προστασία ώστε τα άτομα να μπορούν να ζήσουν σε αξιοπρέπεια. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε για ισορροπία, θα δώσουμε λίγα λεφτά για να έχουμε ισορροπία. Πρέπει να είναι αρκετά για να βρούμε να έχουν τη δυνατότητα αξιοπρέπεια. Η ισορροπία πρέπει να ζητηθεί έναντι των πλουσίων. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποια ελάχιστα εισοδήματα. Η κυρία Τιπούπο. Για τα τρία αυτά σημεία είναι δύσκολο να απαντήσω σε ένα λεπτό. Καταρχήν, εάν υπάρξει η ανάπτυξη θα ακολουθήσουν τα άλλα. Όχι, δεν είναι έτσι. Οι τομεί οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ένδια ξέρουν ότι παρά την οικονομική ανάπτυξη δεν μειώσαμε τι διακρίσει και την ένδια. Θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Να εξασφαλίσουμε ότι θα εργαστούμε για ένα αξιοπρεπέ ελάχιστο ήδη από τώρα ακόμα και σε καιρού κρίση. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ίδια την οδηγία, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν 24 από τι 27 χώρε που έχουν κάτι το οποίο μοιάζει με ελάχιστο εισόδημα. Υπάρχει αυτό. Τώρα σε τρεις χώρες δεν υπάρχει απολύτως τίποτα ή κάτι το οποίο δεν είναι επαρκές. Η κατι το οποιο δεν ειναι επαρκε η Ελλάδα και η Ιταλία. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ήδη <clears throat> μια μορφή συνένεση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως θα πρέπει να εργαστούμε να περάσουμε την ιδέα του ελάχιστου εισοδήματος για τα άτομα ακριβώς που δεν έχουν καμία εργασία, να μπορέσουν να καταρτιστούν καλύτερα, όπω ζητάει η έννοια τη ευέλικτη ασφάλεια, να μπορέσουν να μετακινηθούν κάπου αλλού για να βρουν εργασία, να έχουν τη δυνατότητα να καταναλώνουν, γιατί βλέπουμε ότι στι ΗΠΑ σε εποχή κρίση δίνονται χρήματα σε στρώματα του πληθυσμού που δεν θα τα αποταμιεύσουν, αλλά θα τα καταναλώσουν, θα επανέλθουν στην οικονομία. Όλα αυτά είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστώ που ήμουν τόσο αυστηρή με τη χρήση του χρόνου. αλλά δεν μπορούμε να λαστιχεύουμε το χρόνο στο διενεκές. Κυρία Φίγκερέδο, σας δίνω το λόγο, απλώς υπογραμμίζω τη σημασία και την επικαιρότητα της ε, σημερινής συζήτησης, όχι μονάχα λόγω του πλαισίου κρίσης στο οποίο βρισκόμαστε, αλλά επίσης και γιατί θα πρέπει να αποδεθούμε σε μια πολιτική μάχη γύρω από την έκθεσή σας, γνωρίζοντας ότι η στρατηγική του 2020 έχει σαν στόχο της, με ένα από πέντε στόχους, τη μείωση της ένδυας. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν είναι η επαρκής η προσπάθεια που προβλέπεται να γίνει εκεί. Έχουμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ακοφίν που έλαβε χώρα χθε και που είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Γιατί σε ό,τι αφορά το στόχο της ένδυας, σας διαβάζω στα αγγλικά την παράγραφο που αφορά τα συμπεράσματα, η οποία ουσιαστικά απορρίπτει το στόχο της επίτευξης της εξάλληψη της φτώχειας όπως είχε διατυπωθεί, λέει ότι περαιτέρω εξέταση θα πρέπει να δοθεί στην αρχή και στον σχεδιασμό μιας ενός ενδεχόμενου στόχου κοινωνικής συμπερίληψης ή ένταξης. Ακριβώς τη στιγμή που τα στοιχεία για την ανεργία δείχνουν την επιδείνωση, μια προσέγγιση του ΕΚΟΦΗΝ που δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με τους υπουργού ε, κοινωνικών θεμάτων είναι μια αντιμετώπιση πολύ ανησυχητική και αυτό ίσως θα πρέπει να το λάβει υπόψη η έκθεσή σας. Σας δίνω το λόγο για να κλείσετε αυτή τη συζήτηση κυρία Φιγεϊρέντου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια δύσκολη πολιτική μάχη και όλοι το ξέρουμε. Ορισμένοι από τους παρόντες πριν από χρόνια βρέθηκαν στο πλευρό μου σε μια ανάλογη μάχη τη στρατηγική της Λισαβόνας όταν θελήσαμε τότε να το διαμορφώσουμε αυτό το πρώτο πρόγραμμα της Λισαβόνας. Τώρα ε, είμαστε εδώ σε μια νέα μάχη. Και πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη μάχη παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποια διδάγματα τα οποία αντλήσαμε από όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα και γιατί υπήρξαν και ορισμένα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα καταγράψουμε που είναι η δυνατότητα των φορέων να συναντιούνται μεταξύ τους, να έχουν μια μεγαλύτερη ακτινοβολία έναντι του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τουλάχιστον δυστυχώς το της αγνοεί ακόμα το Συμβούλιο, όπως πολύ σωστά η πρόεδρος μας ανέφερε, γιατί είναι ανάγλυφο αυτό στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Επομένως χρειάζεται να γίνει ακόμα μια πολύ σκληρή και δύσκολη μάχη και χωρίς να επαναλαμβάνω αυτά τα οποία ελέγχθη, σαν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, προτάσεις σας. Σας ευχαριστώ όλους για αυτά τα οποία μας είπατε και αυτά που θα μας δώσετε εγγράφος. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το αδύνατο για να εξασφαλίσουμε τη συνένεση στα θέματα αυτά που είναι τόσο δύσκολα από τη φύση τους, γιατί δεν αρκούν οι δηλώσεις. Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε πολιτικές, πολιτικές νομισματικές, μακροοικονομικής, και ξέρουμε ότι σε όλα αυτά τα θέματα η στάση του Συμβουλίου είναι πάρα πολύ αρνητική. Αν συνεχίσει αυτή η πολιτική, δηλαδή ο μόνος στόχος είναι να μειωθεί στα 3% το έλλειμμα του προπολογισμού των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2013, σίγουρα θα μπορέσουμε να μειώσουμε την ένδια. Γι' αυτό θα πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών είναι μεν σημαντική, αλλά πιο σημαντική από τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών είναι η βιωσιμότητα των κοινωνιών μας, των ανθρώπων που ζουν στις κοινωνίες μας. Δεν είναι αποδεκτό να αυξάνουμε συνέχεια την ένδυα με τις πολλαπλές μορφές της και αιτίες της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός πρέπει να είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο θα πρέπει να οικοδομηθεί αυτή η έκθεση. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες φυσικά να τα συζητήσουμε όλα αυτά για να έχουμε μια ενδελεχέστερη συζήτηση. Για μένα το σημαντικότερο θέμα είναι ακριβώς αυτό το θέμα της βιωσιμότητας της κοινωνίας είναι σημαντικότερο από την εξυγίανση και τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν τα σημεία της συνένεσης. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αποκλείσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Συγγήτρια. Χάρη στο σχέδιο εκθεσή σα. θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ξανά απόψει στι 27 Απριλίου και εν συνεχεία θα δούμε ποια θα είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Τηλεγραφικά θα πάμε στο σημείο 19 και θα το ξεπετάξουμε. Θα σα παρουσιάσω μια, ε, ένα σχέδιο εκνομοδότηση για την εταιρική και κοινωνική ευθύνη σε διεθνεί εμπορικέ συμφωνίε. Πρόκειται για ένα σχέδιο γνωμοδότηση ε, που απευθύνεται στην Επιτροπή ΙΝΤΑ Διεθνού Εμπορίου, που κανονικά θα γινόταν, ε, είχαμε σκεφτεί να ήταν αρχικά επιστολή, αλλά τελικά πήρε αυτή τη μορφή. Ξέρετε τα, το πλαίσιο της γνωμοδότησης, το πλαίσιο στο οποίο κινείται μια γνωμοδότηση. Ε, μην σας εκπλήξει αν ε, υπομορφή τροπολογιών επιμικίνω τον κατάλογο προτάσεων που θα ακούσετε σήμερα. Τώρα, για τη δική μας την Επιτροπή. Η έννοια της εταιρική ευθύνη είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η αιχμή του δόρατος οι εταιρείε. σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους να προωθούν κάποια πράγματα στα οποία βασίζονται οι κοινωνίες μας. Ε, θα πρέπει να υπάρξει κοινωνικός διάλογος ε, όλων των διαφερομένων. Θα γίνει μια συζήτηση ούτως ή άλλως μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων για να δούμε αν η έννοια της εταιρική και κοινωνικής ευθύνης μπορεί να πάρει μορφή νομοθετική ή αν εξορισμού μπορεί να γίνει μόνο να λάβει μορφή μόνο εθελοντική. Επίσης, επειδή μιλάμε για το διεθνές ε, πλαίσιο, ε, έχουμε τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε και τη φοροδιαφυγή και την μαύρη εργασία. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να επαληθεύσουμε ότι δικές μας επιχειρήσεις στο εξωτερικό συμπεριφέρονται υπεύθυνα σε σχέση με τις αξίες που εφαρμόζουν στο εσωτερικό. Δηλαδή, τις ίδιες να εφαρμόζουν και προς τα έξω και στο εξωτερικό. Όταν εξετάσουμε την έκθεση Ορί θα επαληθεύσουμε πώς αυτή η έννοια εντάσσεται στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Νομίζω ότι θα είναι ένας τρόπος για να συνδέσουμε αυτή την έκθεση της Επιτροπής ΙΝΤΑ και την στρατηγική του 2020. Αυτά είναι λίγα στοιχεία που σας δίνω για να δώσω την ακτή μας στη συζήτηση και σας προτείνω τώρα να πάρετε το λόγο. Καταρχάς, δίνω το λόγο στην κυρία Σεσίλια Βίκστρομ ε, από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πρώτη φορά που ως αναπληρωματικά συμμετέχω στην Επιτροπή σας, αλλά επειδή ακριβώς είναι πρώτη φορά θα τα πω στα σουηδικά. Αν θέλετε καμία γλωσσική εμπειρία μη βάλετε τα ακουστικά, αλλιώς βάλτε τα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγεσία για αυτή την ενδιαφέρουσα έκθεση που αφορά ολόκληρη την κοινωνία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, άτομα, πρόσωπα κλπ πρέπει τα νομοσχέδιά μας πάντοτε να εμπεριέχουν την έννοια της κοινωνικής ευθύνης γιατί παρακαλώ μιλώνει την συνέχεια οι συνάδελφοι και δεν μπορώ ούτε ίδια να ακουστώ από τον εαυτό μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρετε, αυτά είναι δύσκολα. Λοιπόν, δεν είναι πρόβλημα, όχι, όχι. Μετά, Λοιπόν, πού ήμουνα, ε, συνεχίζω. Γνωρίζουμε, όπως έλεγα, ότι μπορεί να βελτιωθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, αλλά δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε για την κοινωνική υπευθυνότητα. Αυτό θα, θα έκανε τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα για τις επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να νομοθετήσει για την κοινωνική ευθύνη λοιπόν. Αναφέρομαι στο σημείο 4 ιδιαίτερα όπου γίνεται λόγος για μέτρα που παίρνουν οι επιχειρήσεις και που πρέπει να συμβαδίζουν με την ισχύουσα νομοθεσία ή για το σημείο όπου γίνεται λόγος για δεσμευτική νομοθεσία που να υποχρεώνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να σέβονται την κοινωνική ευθύνη επιχειρήσει τουλάχιστον που συνεργάζονται με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο ρόλος του κράτους εδώ πρέπει να είναι περιορισμένος και να μην υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να ξεπερνούν ακόμη και αυτά που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία στο κράτος μέλος τους. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε την κοινωνική μεν ευθύνη, αλλά οι ελεύθερες συναλλαγές να είναι ο κανόνας και όχι η εφαρμογή δεσμευτικών και προστατευτικών μέτρων. Ο Φρίντμαν και άλλοι αναφέρουν τέτοιου είδους εργαλεία που προσπαθούν οι χώρες μέλη som det är svårt att införa helt och που προσπαθούν μερικές φορές οι χώρες μέλη να εφαρμόσουν. Γιατί δεν μπορεί κανείς να ζητάει την εφαρμογή συνθήκων εργασίας 100% ασφαλών. Γιατί έτσι καταλήγουμε σε διαμάχες των μεν με τους δε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συμμετοχή σας. Δίνω το λόγο σε δύο μιλητές και μετά στην Κομισιόν. Δύο λεπτά ο καθένας. Χάουιτ και Θέρκας. Χάουιτ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να πάρω χρόνο μιλίας από το θέμα μου το οποίο είναι το επόμενο. Εγώ σας ευχαριστώ για την έμφαση που έχετε δώσει στα θέματα της εταιρική κοινωνικής ευθύνης. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή είναι μια έκθεση που έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει τα θέματα της κοινωνικής ευθύνης. Και είναι σημαντικά αυτά που λέγονται στην παράγραφο 5 αυτά μπορούν να αντανακλώνται καλύτερα και στην αιτιολογική σκέψη α σε σχέση με τις ε, δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα στα, στα αγγλικά που λέει ότι δεν πρέπει να σεβόμαστε τα άτομα, απλώ πρέπει να τα βοηθάμε. Αυτό ίσω είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρόβλημα μετάφραση, γιατί υπάρχει συμβατική υποχρέωση να υπάρχει αρρωγή προ τα άτομα αυτά. Σε ό,τι αφορά τώρα τι τροπολογίε, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα των, ε, τα εμπορικά. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικέ οι προτάσει οι οποίε έχουν δοθεί για τι πολυεθνικέ εταιρείε που περιλαμβάνουν ελάχιστα πρότυπα. Πιστεύω θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια πρότυπα στι εμπορικέ συμφωνίε. θα πρέπει να προσαρτώνται σε οποιαδήποτε μορφή αρρωγή που γίνεται για την συνεργασία υπό τη μορφή επενδυτικών συμφωνιών και ρυθμίσεων. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε επίση ότι μέσα στα πλαίσια των κατευθυντηριών γραμμών του ΟΣΑ υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει καλύτερα το πλαίσιο συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι απαραίτητο λοιπόν όλα αυτά τα οποία γίνονται να γίνονται σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά λοιπόν σα τα λέω γιατί δεν έχω πραγματικά χρόνο να αναπτύξω όλα τα θέματα που με ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ ο κ. Σέρκα και ο κ. Κομφεράτη. Εγώ πήρα το λόγο γιατί λένε κάποιοι ότι δεν μπορούμε να νομοθετούμε επιορισμένων ιδεών. Όχι, μπορούμε για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει και έχουμε ήδη νομοθετήσει. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα καταθέσω μια τροπολογία στην εκθεσή σα για να τονίσω ότι η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υποχρέωση που έχουν να σέβονται τις διεθνείς συμβάσεις, ιδίως όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας σε ό,τι αφορά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την ευθύνη τους έναντι των εργαζομένων. Δηλαδή η κοινωνική εταιρική ευθύνη μπορεί να είναι κάτι επιπλέον, μπορεί να είναι το κερασάκι στην τούρτα, κάτι παραπάνω που προστίθεται στις υποχρεώσεις των εταιριών, αλλά δεν απομειώνει τις άλλες τις υποχρεώσεις τους, γιατί αν το κάνει αυτό το πράγμα σημαίνει ότι θα αποδυναμώσουμε τελείως όλο το πλαίσιο της νομοθεσίας που ισχύει για τον χώρο των επιχειρήσεων. κ. Κομφεράτη και μετά η Ευχαριστώ. Η δουλειά που πρέπει να κάνετε είναι, που κάνετε μάλλον, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ειδικά για αυτό το σημείο που, που συζητάμε. Γιατί μέχρι στιγμής η κοινωνική ευθύνη ήταν ε, στην επιλογή και τη διακριτική ευχαίρεια των επιχειρήσεων. Ε, και το διακύβευμα για τι επιχειρήσει ήταν μόνο η αξιοπιστία του, τίποτα άλλο. Εγώ νομίζω όμω ότι είναι απαραίτητο, όχι μόνο δυνατό, να υπάρχουν και δεσμεύσει. Ε, δεν αρκεί η φήμη. Είδαμε τα τελευταία χρόνια επιχειρήσει οι οποίε ε, ε, διένυμαν τεστ για την κοινωνική τους ευθύνη, ενώ την ίδια χρονική στιγμή μόλυναν τη Βόρεια Θάλασσα γιατί επέτρεπαν σε πετρελοφόρα σκουπι, πλοία σκουπίδια να ταξιδεύουν. Ε, και επίσης είχαν εργαζόμενους από χώρες που δουλεύουν ωραιότατα οι ανήλικοι. Νομίζω ότι Αυτή η κοινωνική ευθύνη δεν μπορεί να αφαιθεί στους μηχανισμούς που είχαμε μέχρι εδώ. Πρέπει να δούμε τα πρότυπα, τα κατόφλια και πρέπει και μέσω της συμμετοχής των stakeholders να δούμε ποιες είναι οι δεσμευτικές μορφές ε, που θα επιβάλλουν σε επιχειρήσεις αυτά τα πράγματα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, η κυρία Μπέρτ. Δεν έχετε περισσότερο χρόνο τους βουλευτές, ε. υπόψη, δύο λεπτά κι εσείς. Ευχαριστώ. Από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Να διατρέξω τα σημεία που ακούστηκαν και να δώσω και μία-δύο διευκρινήσει από την ε, Κομισιόν. Καταρχάς, ο ορισμό σα. για την κοινωνική και εταιρική ευθύνη. Στο Α λέτε ότι η ευθύνη ε, είναι τον. Ε, των επιχειρήσεων όπου εθελοντικά ε, ενσωματώνουν κάποια στοιχεία, ε, αναλαμβάνουν κάποιες υποχρεώσεις. Στο σημείο Δέλτα μιλάτε για την αθλητή εργασία και τη φοροαποφυγή. Αυτά είναι παράνομα πράγματα, ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως είναι παράνομα. Ως τέτοια τα βλέπουμε. Επομένω, η κοινωνική και εταιρική ευθύνη δεν, είναι, δεν μπαίνει εδώ. Έπειτα νέα θέματα, κοινωνική ένταξη, α, κάποια ελάχιστα πρότυπα κτλ. Φαντάζομαι ότι μιλάτε για εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ούτω ή άλλω στο εσωτερικό τη ε, Ευρωπαϊ... Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν αυτά τα πράγματα ούτω ή άλλω. Στο σημείο 4 ε, θέλετε ε, αυτή η ευθύνη να επιβεβαιωθεί και νομοθετικά. Εμείς δεν προβλέπουμε σχετικό, σχετική πρόταση νομοθεσίας για το εγγύς μέλλον. Σημείο 6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων ε, με επικοδομητικός ρόλος ό,τι αφορά τις ε, βέλτιστες για την εταιρική ευθύνη. Ναι, βεβαίως, έχει εμπλακεί αυτό το Συμβούλιο στις καλές πρακτικές, αλλά δεν είναι το μόνο το οποίο παράγει τέτοιες ε, βέλτιστες πρακτικές. Από ό,τι ξέρουμε υπάρχουν ε, και άλλα ε, Συμβούλοι Εργαζομένων που εμπλέκονται. Το σημείο 7, πιο δεσμευτικοί κανόνες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε όλο το μήκος αλυσίδας και στους, μέχρι και τους υπεργολάβους. Η Κομισιόν ε, ασχολείται με τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών. Το να ζητήσουμε δεσμευτικούς κανόνες ε, στις εμπορικές συμφωνίες δεν έχει νόημα. Η Κομισιόν δεν είναι σε θέση επίσης να προτείνει νομοθεσία. Αυτά. Ευχαριστώ. Ε, δύο, λεπτά για να δύο λεπτά για να απαντήσετε. Η γνωμοδότηση αυτή είναι μια γνωμοδότηση που αφορά τα θέματα εμπορίου. Αλλά οι πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτούν και κέρδη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή και εκεί συμπεριφέρονται με έναν τρόπο ο οποίος αφήνει πολλά να επιθυμηθούν. Για το θέμα της αδίλωτης εργασίας και της φοροδιαφυγής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει φυσικά μια νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται. Όταν όμως στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν τέτοια πράγματα οι επιχειρήσεις αυτές, εκεί εμπλέκεται και η κοινωνική, του, κοινωνική τους ευθύνη. Είναι μια έγκυρη έννοια εγώ βλέπω άτομα τα οποία έρχονται στο γραφείο μου και μου λένε τι κάνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όταν εξορίσουν μεταλλεύματα στην ΑΒ χώρα ή αναπτύσσουν δραστηριότητες βιομηχανικές παραβιάζοντας όλους τους κανόνες που είναι υποχρεωμένες να σέβονται μέσα στην Ευρώπη. θέτε το θέμα λοιπόν αυτό του διεθνού δικαίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα αντιμετωπίσουμε αυτά με την έκθεση Howard σε λίγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι του εξωτερικού χώρου κάνει μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθούν τα πρότυπα τα οποία έχουμε μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο για κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Το να ζητάμε από τους άλλους να εφαρμόζουν αυτές τις έννοιες και να δεχόμαστε δικές μας επιχειρήσεις όταν βγαίνουν έξω από την Ευρώπη να είναι σκύλοι αλέστε αυτό δεν μπορούμε να το απορρεχτούμε. Πού είναι λοιπόν οι ευρωπαϊκοί, Πού είναι λοιπόν η ευρωπαϊκή, πού είναι η, η, η η ευθύνη των επιχειρήσεων και πού είναι οι νομοθετικές ε, ρυθμίσεις. Εγώ είχα την ευκαιρία να ρωτήσω τους εκπροσώπους της Κομισιόν, αλλά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων σαν ένα επιχείρημα που ουσιαστικά αυξάνει το κύρος μιας επιχείρησης. Παράδειγμα η Total. Όταν η Total λειτουργούσε στην Βυρμανία, έκανε τεράστιες καμπάνιες ε, ε, πληροφόρηση για να δείξει ότι σε, σεβόταν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενώ στη Βερμανία φυσικά δεν ισχύει δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε συνεκτικοί και συνεπεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αυτό είναι μια ελάχιστη μα ευθύνη ω νομοθέτη να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να έχουμε δύο συζητήσει: μία για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και παράλληλα μία για την διακυβέρνηση των επιχειρήσεων. Στον τομέα των επιχειρήσεων θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη των νομοθετικών μέτρων. Αυτό είναι λοιπόν μια συζήτηση που θα έχουμε την ευκαιρία να την αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, απλώ προσθέτω το εξή σε σχέση με το αν το εμπόριο αφορά τι διακρατικέ συμφωνίε. Όχι, υπάρχει και όλα, υπάρχουν όλα αυτά τα διακυβευόμενα όταν πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν τον τζίρο τους ή τα κέρδη τους εκεί που έχουν την έδρα τους και προσπαθούν να αποφύγουν την φορολογία εκεί όπου έχουν καταλυστεύσει τους εθνικούς πόρους χωρών όπου λειτουργούν. Αυτό δεν είναι εμπορικό θέμα. Λοιπόν, σας ζητώ συγγνώμη που είμαι τόσο σύντομη. Αυτό το οποίο σας προτείνω είναι να, κλείσουμε, να σταματήσουμε εδώ τη συζήτηση για αυτό το θέμα σήμερα. Θα επανέλθουμε με την ευκαιρία τη συζήτηση για τις τροπολογίες οι τροπολογίες έχουν χρόνο μέχρι τις 26 Μαρτίου το μεσημέρι να κατατεθούν και στις 27 Μαρτίου θα τις, μάλλον ένα μήνα αργότερα, στις 27 Απριλίου θα τις συζητήσουμε και θα τις ψηφίσουμε στις 28 Απριλίου. Τελευταίο και λουκούμιο σημείο της ημερήσιας διάταξης και δίνω το λόγο στον κύριο Ρίτσαρτ Χάουιτ για να παρουσιάσει την εκθεσή του που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα κοινωνικά περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. 34 τροπολογίες έχουν κατέθει για την εκθέση σας κύριε Χάουιτ και αδειμόνως περιμένουμε την ε, πληροφόρησή σας για αυτές τις τροπολογίες. Έχετε το λόγο κύριε Χάουιτ. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω και εγώ ότι δεν έχουμε πολύ ώρα, γι' αυτό θα τα πω συμπυκνωμένα για να ακούσουμε κυρίως όσους κατέθεσαν ντροπολογίες. Λοιπόν, προσπάθησα στην διατύπωση να διορθώσω τα πράγματα. Κάθε φορά που υπήρχε μια συγκεκριμένη ιδέα, την κράτησα βέβαια. χωρίς να αλλάξει η αρχή του προηγουμένου κειμένου για το θέμα των υπερακτίων εταιριών και άλλα παραδείγματα. Η μόνη τροπολογία που νομίζω ότι θα μπορούσε να συζητηθεί περαιτέρω είναι η δική μου πέντε. 25 Αλλά θα ήθελα να πω στους συντάκτες τα εξής. Ο κύριο Κάπμαν καταρχήν. Η τροπολογία του δεν κάλυπτει ένα θέμα που το είχα αρχικά συμπεριλάβει. Και η 24 μου νομίζω καλύπτει τη δική του, ελπίζω να συμφωνήσει αλλά με απογοητεύουν οι 5, 15, 20 και γιατί είναι δύσκολο εκεί να βρεθεί συμβιβασμό. Για την 5 η, ο ίσος τονισμό στην πρόσβαση και την ανάπτυξη δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Για την 29 μα ακριβώς αυτό είναι θέμα συνδυασμού ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας όπως είπε και ο ΠΟΕ, όπως είπε λέω και ο ΠΟΕ, είναι δύσκολο να συνδυαστούν όλα αυτά. Στον κύριο Ντίκενς θα ήθελα να πω ότι η θέση του στηρίζεται ίσως από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο καταλληλότερος τόπος να τα βάλουμε όλα αυτά. Δεν θέλω να νομίζει ότι είμαι κατά, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι δεν είναι εκτός θέματος. Τον κύριο Χάρκεν τώρα θα ήθελα να μετριαστεί κάπως η διατύπωση, η γλώσσα της τροπολογίας του για να συμφωνεί περισσότερο με τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά δεν είμαι κατά των τροπολογιών του. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ συνοπτικό, κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, κύριε Χάουιτ, για την ε, θαυμάσια γνωμοδότηση. Συμφωνώ ότι κάποιες αντιστροπολογίε σα, ειδικά οι 25, ουσιαστικά λέει τα πράγματα έτσι πιο έντονα, γιατί συχνά η γλώσσα που ε, χρησιμοποιούμε είναι ευχολόγιο. Εσείς πήγατε παραπέρα. Για τις δικές σας τροπολογίες, λοιπόν, μπορώ να τις υποστηρίξω σχεδόν όλες, αν όχι όλες. Ελπίζω και εσείς να υποστηρίξετε κάποιες από τις δικές μου, ιδίω για την ευρύτερη ε, περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Ε, αφορούν την παράγραφο 5. Τώρα, η γνώμη σας ε, ποια είναι για την ε, τροπολογία μου για την παράγραφο 6. Δεν συμφωνούν όλοι. Δεν ξέρω αν την έχετε κοιτάξει. Μπορεί να την κοιτάξετε και αργότερα. Αλλά νομίζω ότι με τις περισσότερες τροπολογίες θα συμφωνήσω. ιδίω με την 32 και την 29. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρη τι επιδιώκουν αυτές τις τροπολογίες. Θα ήθελα οι συντάκτε αν είναι εδώ, να μου εξηγήσουν τι προσπαθούν να επιχειρήσουν αυτέ τι τροπολογίε, γιατί δεν είμαι απόλυτα σίγουρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Higgins. Ευχαριστώ σύντομα, λόγω χρόνου. Αφήνω το θέμα της Κολομβίας. Το έχουμε ήδη συζητήσει εκτενώς. Ένα θέμα, ένα άλλο θέμα που αφορά την επαλήθευση του εάν και κατά πόσον οι επιχειρήσεις πληρούν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ε, πρότυπα που ισχυρίζονται ότι τηρούν. Αυτό είναι πάντα επίμαχο θέμα, γιατί κατ' επανάληψη ε, διάφοροι εκπρόσωποι διαφόρων κοινοτήτων και εργαζομένων έρχονται, προέρχονται από χώρες ε, και σε εταίροι των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρνουν στοιχεία με αποδείξεις για το αντίθετο. Ε, εν συνεχεία οι επιχειρήσεις βέβαια το αρνούνται αυτό. Το θέμα λοιπόν να υπάρξει επαλήθευση του κατά πόσον ατύρουν αυτά τα πρότυπα. Ο κύριος ε, Χάουιτ προσπαθεί να το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα στην παράγραφο 8 με ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη για τη συμμόρφωση των ε, εταιριών και τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούν. Ε, πρέπει οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις διαφόρων κοινοτήτων που είναι τα πρώτα θύματα των προβλημάτων που δημιουργούν οι επιχειρήσεις να εμπλέκονται στην εξέταση των όποιων παραπώνων και στη διεκπαιρέωση αυτών των ε, αγωγών, ας πούμε. Αυτά ευχαριστώ. Λίγα σχόλια. Δεν θα επαναλάβω αυτά που, κάναμε, αυτά που είπαμε προηγουμένω. Λέει εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την γνωμοδότηση. Ε, χαιρόμαστε που εμπλέκεται η Επιτροπή Απασχόληση. Διάφορε ανησυχίε που εκφράσαμε ισχύουν και εδώ, ειδικά ε, σε ορισμένε παραπομπέ σε άρθρα του ΠΟΕ. Θα ήθελα να θίξω ένα-δύο σημεία στις τροπολογίες της παραγράφου 3, εκεί όπου μιλάμε για την διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών. Θα προτιμούσαμε να μιλήσουμε για τους κοινωνικούς εταίρους εκεί και όχι για τους stakeholders, όχι για τους ενδιαφερόμενους. Να συμπεριλάβουμε και τα συνδικάτα, αλλά και όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Έτσι, για την 5, το ξαναείπαμε, θα το ξαναπώ και τώρα. Είναι μια γενική γνωμοδότηση για την εμπορική πολιτική. Δεν νομίζουμε ότι είναι σκόπιμο να αναφερθούμε σε ειδικέ περιπτώσεις ή ειδικέ χώρες. Κάθε μία από αυτές θα πρέπει να εξεταστεί εξατομικευμένα ανάλογα με τα προβλήματα και τα θετικά του στοιχεία. Καλό θα ήταν να σβήσετε τις αναφορές σε οποιασδήποτε χώρες έχετε. Ένα-δύο σχόλια τώρα. για τις κατευθυντήριες γραμμές και τον, την προαιρετική φύση των κατευθυντήριων γραμμών του ΩΣΑ. Για τις τροπο... Προτιμώ την τροπολογία 24 που μιλάει για την, ε, το να υπόψη της τι ε, γραμμές. Παράγραφος 7. Έτσι. Τώρα, παράγραφος 8. Αντί να μιλάμε για τις αποφάσεις των ανεξάρτων ε, πυρογνωμόνων, να μην μιλάμε ε, για αποφάσεις, αλλά για εκθέσεις, γιατί τις αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι πυρογνώμονε, τις παίρνουν τα κράτη. Είναι πιο σωστό όρο. Ο κ. Κάσλι δεν είναι εδώ δυστυχώ, άρα δεν μπορεί να μιλήσει για την τροπολογία του 29 και 32. Αλλά νομίζω ότι σχετίζονται με αυτά που είπε η Κομισιόν και προηγουμένω. Ε, δηλαδή η συμμόρφωση με τα διεθνή εργατικά πρότυπα δεν συνδέονται μόνο με τον Mode 4 ή με τις υπηρεσίες. Πρόκειται για πρότυπα που ισχύουν γενικά. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να βγάλετε ίσως την παράγραφο 9. Τώρα, παράγραφος 10 ορισμός της επιδότησης των ΠΟΕ ε, ούτως ή άλλως εναρμονίζεται με τις δικές μας, με τους δικούς μας ορισμούς. Ε, δεν υπάρχει λόγος να τα αλλάξουμε. Ε, τώρα, για την απασχόληση των ανηλίκων ε, του Τόμας Μαν. Πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε ένα έγγραφο εργασίας για αυτό το θέμα ε, και η σας Επιτροπή είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή για το θέμα αυτό. Ίσως λοιπόν θα ήταν ε, καλύτερο το σημείο αυτό να το λάβετε υπόψη σας στη συζήτηση που θα κάνετε για το έγγραφο του προσωπικού της Κομισιόν. Ευχαριστώ ο εισηγητής. Thank you. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Χάρκιν μου ζήτησε να δω την τροπολογία της στην υπαριθμό 17. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να αναφερθούν ε, τα εργασιακά πρότυπα. Για τα θέματα της Λατινικής Αμερικής άκουσε αυτό που λέει δηλαδή η Κομισιόν που λέει δεν θέλει να αναφέρεται ειδικά οποιαδήποτε χώρα. Προφανώς αναπόκειται στο Κοινοβούλιο να αποφασίσει αν θέλει να αναφερθεί σε μεμονωμένες χώρες ή όχι. Δεν είναι θέμα της Κομισιόν. Αυτό το οποίο θέλω να πω στην κυρία Χάρκιν και στην Επιτροπή όμως, στην Κομισιόν, ότι εγώ προσπάθησα να είμαι πάρα πολύ προσεκτικό στη σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης για να μην πω ότι είναι καλές ή κακές συμφωνίες για την παιδική εργασία με ορισμένες χώρες. Γι' αυτό εγώ υποστήριζω τη δική μου τροπολογία. Γιατί δεν είναι εδώ το σημείο που θα επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά για τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στα πλαίσια της αξιολόγησης για τη βιωσιμότητα που αναφέρει και η κυρία Χάρκιν, η Κομισιόν έχει κάνει κάποιες μνήες αυτών των χωρών. Και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πω ότι δεν έχει το δικαίωμα η Κομισιόν να άρει αυτές τις μνήες σε τέτοιες χώρες. Ίσως με την κυρία Άρκιν να τα βρούμε μετά από την συνεδρίαση αυτή για τη συγκεκριμένη διατύπωση που αφορά τη Λατινική Αμερική. Θέλω να είμαι απόλυτα επακριβής σε σχέση με τα πραγματικά στοιχεία για τους λόγους που ανέφερε και η Κομισιόν, αλλά δεν είμαι εναντίον αυτής της ε, πρότασης της κυρίας Χάρκιν, απλώς θέλω να βρούμε την καλύτερη διατύπωση για αυτά που είπε ο κύριος Higgins για την επαληθευσιμότητα. Συμφωνώ απόλυτα, οι τροπολογίε του και οι δικέ μου τροπολογίε είναι απόλυτα συμβατέ. Ελπίζω λοιπόν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία εποφελή συμβαστική λύση. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι. Εγώ έχω εξετάσει μια τροπολογία ενός μέλους που δεν είναι παρόντες εδώ αλλά η άποψή μου εδώ εξετάζει τις διάφορες ερμηνείες οι οποίες μπορούν να υπάρχουν για αυτά τα θέματα. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Μπορεί να πει κάποιος ότι η Κομισιόν συμμερίζεται ή όχι την άποψη του Α ή του Β βουλευτού, αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί να δίνουν μια τελείως διαφορετική άποψη και δεν νομίζω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να είναι αμυντική σε σχέση με τη στάση της. Τώρα, για τους κοινωνικούς εταίρους, αν θέλουν κάποιοι βουλευτές να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, μπορούμε να το κάνουμε. Στη συνέχεια είπα για τις ειδικές χώρες που αναφέρονται. Η Κομισιόν έχει ήδη εκφράσει την άποψή της για τις κατευθυντήρες γραμμές του ΩΣΑ και νομίζω ότι κατανοώ ότι υπήρξε μια αμφισημία στο αρχικό κείμενο. Όταν όμως υποστηρίζουν τις ε, τη ε, τροπολογίες του κ. που δεν θέλουν καμία μνήμα σε σχέση με συμμόρφωση με τα εργασιακά ε, του εργασιακού κανόνε ακόμα και στα πλαίσια του ΠΟΕ αυτή είναι μια αρκετά ακραία θέση είπε ότι υποστηρίζει η Κομισιόν τη Τροπολογία 32 και 29 με 32 αλλά θέλουν να υπάρχει συμμόρφωση με τα εθνικά στάνταρ μέσα από άλλα μέσα δεν λέει αυτό όμως η τροπολογία 34. Γιατί 32 μπορεί η Κομισιόν να μην θέλει την ερμηνεία ή δεν συμφωνεί σήμερα με αυτή. Αλλά αυτή η τροπολογία περιλαμβάνει και το να εξετάσουμε το ρόλο των εργασιακών προτύπων στον ΠΟΕΠ. Άλλοι λένε ότι θα πρέπει να υπάρξει και συγχώνευση του ΠΟΕ με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και να είναι υποχρεωτικά τα πρότυπά του. Εγώ λέω απλώ να δούμε όλε τι πτυχέ τη τροπολογία προτού δεχτείτε το σύνολο τη τροπολογία 32. Αλλά είναι κάπω αργά, είμαστε στο τέλο τη ημέρα και λίγοι καυγάδε ίσω μα βοηθάνε να καταλάβουμε καλύτερα τα θέματα που είναι ενώπιον μα. Ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. Εγώ πάντα είμαι. με. <coughs> Όταν οι προσκεκλημένες επιτροπές παρεμβαίνουν στις, ε, συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προσκαλείται ε, παρεμβαίνει στις ε, συνεδριάσεις μας. δεν μιλάω για τους επιτρόπους, έτσι. Τους καλούμε να συμμετάσχουν στις εργασίες μας ως υπηρεσία από την οποία απορρέει η κάθε νομοθεσία. Ο στόχος της ανταλλαγής αυτής απόψεων, και το λέω και για τις δύο παρεμβάσεις που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι, ο στόχος αυτής της α, παρέμβασης είναι να μας βάλει στο σωστό τεχνικό δρόμο. Να μας μιλήσει για την νομική βάση, για τις προθέσεις της Κομισιόν. Αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι πολιτική αξιολόγηση της άποψης του βουλευτή ή του εισηγητή ή των βουλευτών ε, κατά την συνεισφορά τους ε, για την ε, εκπόνηση των ε, κειμένων πολιτικών ή νομοθετικών. Το λέω για πρώτη φορά με τόσο στεναρό τρόπο. Το λέω και για την, τους συναδέλφους από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΗΝ και για την Γενική Διεύθυνση Απασχόληση. Ο ρόλος της Κομισιόν όταν εμπλέκει εργασίες μας δεν είναι να μας κάνει πολιτική αξιολόγηση για τις δικές μας πολιτικές απόψεις. Τούτου λεχθεντο σας ευχαριστώ για την πραγματογνωμοσύνη σας, η οποία είναι σημαντική. Όχι, δεν σας δίνω τον λόγο, γιατί τελείωσε ο χρόνος, μας. Θα σας συναντήσω μια άλλη φορά. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Και θα υιοθετήσουμε την γνωμοδότηση του κυρίου Χάουιτ στη συνεδρίαση της 28 Απριλίου. Σας δίνω ραντεβού για την επόμενη